Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, θα ήθελα να αρχίσουμε την ημερήσια διάταξη. Είναι ιδιαίτερα μεστό το πρόγραμμά μας σήμερα. Πολλά και διάφορα σημεία για τη συνεδρίασή μας. Γι' αυτό ας εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Αν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις, θα την εγκρίνουμε. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προέδρου. Το σημείο 7 τη ημερήσια διάταξης τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρε, δεν ισχύει το σχέδιο έκθεσης που έχετε λάβει στο ντοσιέ σα. Θα λάβετε ένα νέο σωστό στην επόμενη συνεδρίαση. Έχετε λάβει και τα πρακτικά. Αν έχετε σχόλια, μπορείτε να υποβάλλετε και τα διάφορα τα αιτήματά σας στη γραμματεία. Μην ξεχνάτε ότι η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται απευθείας από το webstream. Γιατί θα συζητήσουμε και κάποια θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μετά την αναδιάρθρωση του Γραφείου συνταξή. η κυρία Τατιάνα Μναζίκοβα. Συγγνώμη που κατακρεώργησα το όνομά σας. Αντικαθιστάτε κυρία Αγνιέσκα Πικάρσκα. Μάλλον όχι. Και η κυρία Πιακάρσκα έρχονται στη γραμματεία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Τα πρακτικά της συνεδρίας των συντονιστών της 10ης Δεκεμβρίου σας έχουν μοιραστεί. Και για τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου τα πρακτικά θα σας τα μοιράσουμε αργότερα. Αν δεν υποβάλλετε στάσεις θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Έγκριση των πρακτικών τώρα της συνεδρίασης της 7ης Δεκεμβρίου και αυτά θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Και πάμε στο πρώτο ουσιαστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 5, επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο παγκόσμιο εμπόριο. Οι συντονιστές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα σχέδιο που θα υποβάλουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε για τη σύνταξη προφορικής ερώτησης. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής ερώτησης. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Οπότε εγκρίνεται η προφορική ερώτηση. Σημείο 6. Εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αρχίζει η ακρόαση μας τώρα. Έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες καλεσμένους Θα σας τους παρουσιάσω. Πρόκειται για τον Δόκτωρ Σαβαλάλα από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ στις κατοχώρες. Είναι λέκτορος του Πανεπιστημίου στη Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και στη θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ όπως σας είπα. Ε, θα σας μοιράσουμε και το βιογραφικό του. Δόκτωρ Χάουαρντ, Διευθυντής ε, του Τμήματος Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ε, της Ομοσπονδίας, Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδικάτων στο Βέλγιο. Μάλιστα, ήταν διευθυντής του τμήματος, είναι διευθυντής του τμήματος κοινωνικών και κοινωνικών υποθέσεων από το 2006. θα σας μοιράσουμε και το δικό του βιογραφικό και τέλος, Dr. Quick. Διευθυντής Εμπορικής Πολιτικής στο VCI, την Ένωση Σωματείο μάλλον ε, Χημικής Βιομηχανίας. Επίσης ήταν αντιπρόεδρος μιας ομάδας εργασίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου και ε, αντιπρόεδρος σε μια ομάδα του, του Business Europe. Ο κύριος Γιου που προβλεπόταν αρχικά ως εμπειρογνώμων στην ακρόαση κολλείεται και δεν θα έρθει. Θα δώσω τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας και μετά στα μέλη της Επιτροπής για ερωτοπαντήσεις. Κάποια διαδικαστικά καταρχήν. Όπως ξέρουμε, οι εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα διεθνούς εμπορίου εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Και διμερείς, ε, ε, επαφές ε, ελεύθερου εμπορίου εντάσσονται σε ένα πλαίσιο γενικότερο και εκτενέστερων εμπορικών συμφωνιών που έχουν και πολιτικό ιστορικό. Υπάρχουν άλλωστε και οι συμφωνίε σύνδεση που κανονικά περιλαμβάνουν και ρήτρε για ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικές προδιαγραφές, αλλά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Είναι γνωστό τη σπάση ότι ε, οι βασικοί εταίροι στην παγκόσμια σκηνή δεν συνδέουν πολλές φορές τις εμπορικές συμφωνίες με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ή τουλάχιστον δεν το κάνουν ε, ε, στο βαθμό που το επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πολλοί προβληματίζονται κατά πόσο η ευρωπαϊκή πολιτική που πρωτοστατεί στην πρόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων ε, μέσω εμπορικών συμφωνιών είναι επιτυχής. Και αν όντως ε, οδηγεί τον κόσμο σε εκτενέστερες εμπορικές συμφωνίες ή μήπως αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την φέρνει σε δυσμενή θέση ε, απέναντι στους εταίρους της, όπως επιχειρηματολογούν κάποιοι άλλοι. Οπότε θα πρέπει να αναλύσουμε κατά πόσο τέτοιου είδους ρήτρε όντως ε, εκπληρούν τους στόχους τους, δηλαδή τη βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ε, συνθήκων στις τρίτες χώρες ή τις ενδιαφερόμενες χώρες ή μήπως έχουν ανεπιθύμητα αρνητικά αποτελέσματα και παρενέργειες. Είναι προφανές ότι για να είναι πιο επιτυχής η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προώθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών της αρχών μέσω των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει και να ε, εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτών των ρητρών και προτύπων από τις τρίτες χώρες που εμπλέκονται σε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Ελπίζω με τη δημόσια αυτή ακρόαση να διαλευκάνουμε κάπως αυτό το πολυσύθετο ζήτημα και να αρχίσουμε και λίγο φως στο ερώτημα το πώς θα βελτιώσουμε την πολιτική μας για να εφαρμόσουμε τις αρχές μας στον τομέα αυτό. Χωρίς άλλη λοιπόν χρονοτριβή, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρώτο μας εμπειρογνώμονα, από τους τρεις που σας ανέφερα τον κύριο Νταλιντιέμπο Σαμπαλάλα το Πανεπιστημίου του Μάστριχτ. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να σεβαστώ το χρόνο σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας μιλήσω για ορισμένο χρόνο που θα ακολουθηθεί από ερωταπαντήσεις. Θα έπρεπε να σας πω ότι πριν εργαστώ στο Πανεπιστήμιο της Μαστρίχτης είχα μια θέση στο Διεθνές κέντρο εμπορικού δικαίου που χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα μη κυβερνητικέ οργανώσεις από και για χώρες ΑΚΕ. Και από εκείνη την εμπειρία με διαπραγματεύσεις από τέτοιες οργανώσεις έχουν προκύψει τα συμπεράσματά μου. Θα περιγράψω και λίγο γενικότερα τα πράγματα, ίσως να τα ξέρουν ορισμένοι από εσά, όχι όμως όλοι σίγουρα αυτά που θα πω. Υπάρχει μεγάλη παράδοση στην Ένωση για τη σύναψη εμπορικών σχέσεων με τις πρώην απικίες της και εδώ συνδυάζονταν πάντοτε, αυτό συνδυαζόταν πάντοτε με τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που είχαν. Οι όλο και περισσότερες συγκεντρωτικές δικαιοδοσίες της Ένωσης, ιδιαίτερα για τα εμπορικά που εκφράζονται από την Κομισιόν, έχουν οδηγήσει στο γεγονός ότι οι εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες αυτές να έχουν διευρυνθεί και σε άλλους εταίρους όχι παραδοσιακούς όπως οι πρώην απικίες. Υπάρχουν οι χώρες πρόσφατης εκβιομηχάνησης και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη πλέον εκτός από τα εμπορικά και περιβαλλοντολογικά και πολιτιστικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι έχει αλλάξει το κέντρο βάρους της διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες αυτές γιατί από σύστημα προτιμήσεων έχουμε περάσει σε ένα σύστημα αμοιβαιότητα από δασμολογικά σε γενικότερα κανονιστικά θέματα και τέλος η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες από αυτές τις δικαιοδοσίες διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι η γενική αυτή διεύθυνση κυρίως ασχολείται εκ μέρους της Επιτροπής με τα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά θέματα. Έχει και ο ΠΟΕ προσπαθήσει να διευθετήσει διεθνώς τέτοια θέματα, αλλά φαίνεται ότι η εξωτερική πολιτική, ιδίω ως προς τα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά, χαρακτηρίζεται από την απροθυμία της Γενικής Αυτής Διεύθυνσης να χορηγήσει δικαιοδοσίες σε άλλους και άλλα εξαρτώνται όλα σχεδόν από τη γενική αυτή διεύθυνση και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη ή έτσι υπάρχει μάλλον λιγότερη συνοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική γιατί μεταφέρονται όλο και περισσότερα στοιχεία στην Γενική αυτή Διεύθυνση. Για να δούμε ποια είναι τα κύρια στοιχεία που πρέπει να συζητήσουμε εδώ, πρέπει να μιλήσουμε και για τους ανταγωνιστές της Ένωσης και κυρίως την Κίνα. Ιδιαίτερα το τι αντιπροσωπεύει η χώρα αυτή για παραδοσιακούς εταίρους της Ένωσης όπως τις Αφρικανικές χώρες. πρέπει να σημειώσουμε ότι οι συμφωνίες, οι καινούργιες αυτές συμφωνίες χαρακτηρίζονται από δύο στοιχεία. Πρώτον, η λεγόμενη no strings attached ιδεολογία και η δεύτερη ότι πρόκειται για νέο, είδο, νέο είδος συμφωνιών που δεν αφορά καθεαυτές εμπορικές συμφωνίες. Άμα δούμε λοιπόν από τι χαρακτηρίζονται οι συμφωνίες αυτές, διαπιστώνουμε ότι το κυριότερο θέμα είναι το κατά πόσον οι συμφωνίες καλύπτουν και τον κοινωνικό, όχι μάλλον τόσο το κατά πόσον καλύπτουν οι συμφωνίες τον κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα, αλλά μάλλον την πρόσβαση στις αγορές. για να δούμε κατά πόσον χρειάζεται να συμπεριληφθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό στοιχείο πρέπει να εξετάσουμε το εξής. Δεν να αποφευχθούν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συμπερίληψη των στοιχείων αυτών στην σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας σήμερα. Γιατί τώρα υπάρχει δυνατότητα το εμπόριο να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία αυτά αυτόματα σχεδόν στις συμφωνίες. Αν δεν τα συμπεριλαμβάνει, τότε έχουμε μια καθαρά μερκαντιλιστική αντίληψη και όχι μια ολοκληρωμένη τι αυτή. Να σας δώσω δύο παραδείγματα από την εμπειρία μου με τέτοιες διαπραγματεύσεις. Το ένα αφορά το εύρος της εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν για την πνευματική διοκτησία. Έχουμε διαπιστώσει ότι παραδείγματος χάρη η Ολλανδία κατέσχεσε φάρμακα τα οποία έχουν παραχθεί νόμιμα στην Ινδία και τη Βραζιλία αλλά έχουν απαγορευτεί για εισαγωγή στην Ένωση. Και οι κυβερνητικές προμήθειες είναι το δεύτερο παράδειγμα. Στη Νότια Αφρική έχουν ληφθεί μέτρα ποσοστώσεων υπέρ επιχειρήσεων μαύρων προϊόντα των οποίων όμως μπορεί να απαγορεύονται να εισαχθούν στις χώρες της Ένωσης. Τέλος. Η Ένωση έχει διεθνείς υποχρεώσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον που είναι υποχρεωμένη να σέβεται και κατά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Αλλά ο αυτόνομος σχεδόν χαρακτήρας του εμπορίου σημαίνει ότι δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Και το πρόβλημα για την Ένωση δεν είναι ότι υπάρχουν οι πτυχές αυτές του εμπορίου αλλά ότι είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν πλήρως ακόμη και στις καθαρά εμπορικές συμφωνίες που πρέπει να συνάψει. Και γι' αυτό έχω εφεύρει την έννοια του doing better αντί doing without που λένε. Για τα κοινωνικά υπάρχουν τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και άλλες συμβάσεις όπως της Βασιλείας. Η Ένωση είναι υποχρεωμένη τουλάχιστον να σέβεται αυτές τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει. Αλλά επιπλέον πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές και εσωτερικά και άρα είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλαμβάνει κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά θέματα και μέτρα κατά τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας. Εδώ βέβαια πρόκειται για ευκαιρίες πληρέστερης εφαρμογής κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών συμφωνιών. Υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες στα πλαίσια του ΠΟΕ και είναι προφανές ότι αυτές επηρεάζουν και ανεξάρτητες περιβαλλοντολογικές ή κοινωνικές συμφωνίες και μέτρα. Αλλά έτσι Δίνεται επίσης η ευκαιρία να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Άλλο συμπέρασμα που έχω βγάλει από την εμπειρία μου με τις διαπραγματεύσεις είναι ότι φαίνεται όλο και μεγαλύτερο το χάσμα μεταξύ αυτών που δηλώνει επισήμως η Ένωση για τα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά και αυτών που όντως προτείνει σε μια διαπραγμάτευση. Αυτόν που είναι διατεθειμένοι δηλαδή να υποστηρίξει πάση θυσία και αυτόν που είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσει. Για τα εμπορικά επιμένει βέβαια, αλλά για τα υπόλοιπα, δηλαδή τα περαιτέρω, τα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά, είναι διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις. Αυτό φυσικά οφείλεται στην κυριαρχία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, αλλά έχει μειωθεί και η αξιοπιστία διεθνώς των πρόσθετων αυτών μέτρων όταν πρόκειται για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων. Και οι άλλες χώρες βλέπουν ότι δεν προσφέρει τίποτε παραπάνω η προσθήκη αυτών των πρόσθετων μέτρων γιατί δεν υπάρχει πια κανένα μονοπόλιο σε αυτά. Επομένως, η Ένωση θα έπρεπε να επιμείνει σε αυτά τα πρόσθετα μέτρα ως κάτι που δίνει μεγαλύτερη αξία ανταγωνιστική έναντι των ανταγωνιστών της δηλαδή. Ευχαριστώ. Α, ευχαριστούμε πολύ για την σαφέστατη αυτή παρουσίαση. Η γραπτή της μορφή έχει κατατεθεί και θα διανεμηθεί εκ των υστέρων. Και τώρα ο κύριος Χαουάρντ από τη Διεθνή Εμπορική Ομοσπονδία του Βελγίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ για εδώ σήμερα. Είμαστε βασισμένοι στο Βέλγιο, αλλά εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους σε 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην παρουσίασή μου θα επικεντρωθώ στα κοινωνικά πρότυπα, επειδή έχουμε και χρονικούς περιορισμούς, αν και φυσικά συμφωνούμε ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα και θέματα θα πρέπει φυσικά να λαμβάνονται και αυτά υπόψη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Να ξεκινήσω αναφέροντας κάποιους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα αυτά και να πούμε και τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διμερές επίπεδο αλλά και σε πολυμερές επίπεδο διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τώρα το γιατί θεωρούμε ότι τα θέματα αυτά είναι σημαντικά. Πριν από 10 χρόνια περίπου υπήρχε μία υπόθεση ότι το εμπόριο ήταν κατοφατικό και άρα δεν υπήρχε λόγος να συζητηθούν θέματα όπως ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως ε, είπε όμως και ο προηγούμενος ομιλητής. Πλέον υπάρχει μία συμφωνία, μία συνένεση ότι υπάρχει αντίκτυπος του εμπορίου στα πρότυπα αυτά. Και αυτό εκφράζεται στην ε, σχετική έκθεση του ILO, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας με, την ε, αποτελεσματική καθοδήγηση του κυρίου Λαμή στον ΠΟΕ έχουν εξευρεθεί διάφοροι τρόποι με, τον οποίο, με τους οποίους ο αντίκτυπος του εμπορίου αποδεικνύεται να μην είναι απαραίτητα θετικός. Αυξάνεται σε πολλές χώρες η ανισότητα, όχι παντού αλλά σε πολλές χώρες και σε πολλές περιπτώσεις αυξάνεται και η αβεβαιότητα της θέσης, των θέσεων εργασίας καθώς αυξάνεται και η κινητικότητα της παραγωγής στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Δεν υπάρχει αυτόματη σχέση μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης, ούτε μεταξύ εμπορίου και της ε, μείωσης της στόχιας. Άρα η έκθεση αυτή είναι σημαντική, θεωρώ, αποτελεί τη βάση για να αναθεωρηθούν κάποιες υποθέσεις, εικασίες για την αυτόματη θετική φύση του εμπορίου. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε και το τι συνέπειες υπάρχουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων από το εμπόριο. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ε, παραβίασης ε, βασικών εργασιακών προτύπων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον τομέα των ε, κομμένων λουγιών. Είναι απαράδεκτες οι ώρες εργασίες, η πίεση που δέχονται τα συνδικάτα η χρήση των φυτοφαρμάκων και των άλλων χημικών για την προώθηση της παραγωγής και το ίδιο ισχύει για πολλούς τομείς πρώτων υλών, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή καπνού και βακιού στην Κεντρική Ασία, όπου χρησιμοποιείται και παιδική εργασία για την αύξηση της παραγωγής, επίσης την παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων, κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης, όπου προκύπτει ένα μοντέλο χαμηλών εισοδημάτων, μισθών για την αύξηση των εξαγωγών και σε ό,τι αφορά τον ε, τομέα μεταποίησης των εξαγωγών που αφορά πάνω από 50 εκατομμύρια εργαζόμενους όπου βλέπουμε ότι η απουσία συνδικάτων είτε λόγω της πίεσης της νομοθεσίας είτε της μεμονωμένης πίεσης που δέχονται και η θυματοποίηση των εργαζομένων σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, είτε προβλήματα υγείας, είτε προβλήματα α, πληρωμής των αμοιβών, είτε έλλειψη κοινωνικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά καταδεικνύουν το μεγάλο φάσμα προβλημάτων που προκύπτουν ουσιαστικά από το εμπόριο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ αναφέρονται τα στοιχεία αυτά και από μονομένες χώρες και ζητείται από μονομένες χώρες αλλά και από το σύνολο των ε, χωρών να διεξάγουν σχετικές μελέτες αντικτύπου με τη χρήση των εμπειρογνωμόνων και της τεχνογνωσίας των μεμονωμένων υπηρεσιών προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να δοθεί μια καλή σύνοψη των ενδεχομένων συνεπειών. Και επίσης μακροπρόθεσμα ένα πρόγραμμα εργασία στα πλαίσια του ΠΟΕ, το οποίο θα καλύπτει αυτό το πολύ βασικό ζήτημα. Ένα πρόγραμμα εργασίας μπορεί να, ξεκινήσει, να ξεκινήσει ανεξάρτητα από την σύναψη και την επιτευξή συμφωνία στα πλαίσια του γύρου τη ΔΟΧΑ. Δεν υπάρχει λόγο να τα συνδυάσουμε αυτά. Θα πρέπει να συνεργαστεί ο ΑΕΛΟ με τον ΠΟΕ για να εξεταστούν τέτοια προβλήματα. Επίσης, μια αλλαγή των θεμάτων σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των πολιτικών σχετικά με το εμπόριο στα πλαίσια του ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει επικοδομητικές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τα πολιτικά αυτά πρότυπα, αλλά αυτό γίνεται ουσιαστικά σε βάση ad hoc. Τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αντιδράση των κυβερνήσεων είναι αρκετά απρόβλεπτα. Πολλέ κυβερνήσει αρνούνται να συζητήσουν τέτοια θέματα, ακόμα και όπου είναι προφανή η σχέση μεταξύ των εμπορικών πολιτικών τους και της κατάστασης των εργασιακών προτύπων στου ανάλογου τομείς εξαγωγών. Και υπάρχουν και άλλοι τομεί τους οποίου ο ΠΟΕ θα μπορούσε να αυξήσει την ε, πολιτική του σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Ξεκίνησε την δεκαετία του 90 μια προσπάθεια, αλλά δεν δόθηκε μεγάλη συνέχεια και θα άξιζε να συζητηθεί το θέμα αυτό περαιτέρω στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Νομίζω ότι προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις για το θέμα αυτό και για να προωθηθεί η ιδέα της αξιοπρεπούς εργασίας παγκοσμίω, θα πρέπει να επιδιωχθούν οι στόχοι αυτοί. Αυτά σε ό,τι αφορά την πολυμερή ατζέντα, όπου θεωρούμε ότι είναι σωστό να συμπεριληφθούν οι παράγοντες περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί. Σε διμερές επίπεδο, και ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα πρέπει να προβούμε σε μια δήλωση την οποία και τη βλέπετε συνημένη σε ό,τι αφορά την δήλωση των συνδικάτων Έχουμε λοιπόν 14 αρχές οι οποίες θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στα κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης στις διμερείς ε, διαπραγματεύσεις της Ένωσης για την ε, ελεύθερο εμπόριο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από δέσμευση και των δύο μέρων να σεβαστούν τα πρότυπα εργασίας και να περάσουμε και στην επικύρωση των οκτώ συμβάσεων του ILO για την εργασία. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τις διμερείς διαπραγματεύσεις. Και όπως είπε ο πρόεδρος Μορέρος στην αρχή, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν επίσης αυτοί οι παράγοντες, αυτές οι συνιστώσεις. Και βλέπουμε ποια είναι η διαφορά με την τρέχουσα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζουμε βέβαια πολλά θέματα από αυτά που αναφέρει για το περιεχόμενο των κεφαλαίων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλυφθεί και δράση για να αποδειχθούν αποτελεσματικά αυτά τα κεφάλαια. Θα πρέπει να υπάρχει και μία σύνδεση με τις σχετικές διατάξεις με το κύριο σώμα των συμφωνιών. Και θα πρέπει να υπάρχουν και διατάξεις υλοποίησης, εκτέλεσης για τα κεφάλαια αυτά. Και αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες διατάξεις των διμερών συμφωνιών. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα θέλαμε να συμπεριληφθεί και το οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση είναι η δέσμευση και των δύο μερών να γίνουν σεβαστά τα πρότυπα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς επιχειρήσεις και δέσμευση ότι τα μέρη δεν πρόκειται να χαμηλώσουν τα πρότυπα εργασίας για να προσελκύσουν επενδύσεις. Θα θέλαμε να υπάρχει διάταξη για την διαρκή αξιολόγηση της βιωσιμότητας των σχέσεων αυτών και θα θέλαμε να υπάρχει και εποπτεία των κοινωνικών εταίρων για να επισημαίνονται περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής παραβίαση των προτύπων εργασίας και των άλλων στοιχείων των συμφωνιών. Αυτά τα θέματα λοιπόν συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και, ε, παράδειγμα στις συμφωνίες με την Κορέα και την Καραϊβική όπου εξετάζουμε τη διαδικασία επικύρωσης για να διασφαλίσουμε ότι όντως αυτοί οι όροι θα τηρηθούν πλήρως. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα θέματα συμμόρφωσης, θα θέλαμε επίσης ε, να υπάρχει κάποια πρόβλεψη όχι μόνο για την απόσυρση των εμπορικών προνομίων, αλλά και ένα νέο μέτρο το οποίο υπάρχει σε κάποιες συμπορικές συμφωνίες να χρησιμοποιούνται ενδεχομένω και πρόστιμα σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι συμφωνίες. Και αυτά τα πρόστιμα θα μπορούσαν να ανακυκλώνονται υπέρ του συμφέροντος της χώρας, να ανταπανηθούν δηλαδή για να βελτιωθούν οι κοινωνικές, ε, τα κοινωνικά πρότυπα στους τομείς όπου δεν υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση. Πρόεδρε, Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ένωσης και όπως σας είπα θεωρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρωτεύοντα ρόλο και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την ε, Κορέα και σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Αλληλείας με την Ινδία, με τις χώρες Ασιαν, της Λατινικής Αμερικής και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει για τη συνεργασία και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων για την ε, αποτελεσματική του υλοποίηση. Ευχαριστώ πολύ, λέω. Ευχαριστούμε για την ε, δήλωσή σας για τη θέση των συνδικάτων ως προς το θέμα αυτό. Ο κύριος Χάουαρτ μα μοίρασε και δύο έγγραφα. in his... Τα ανέφερε και στην ομιλία του για τα αιτήματα σε ό,τι αφορά βασικά και στοιχειώδη κοινωνικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά τα θέματα ανάπτυξης στις ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ένωσης για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Επίσης είχαμε και την 7η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ του περασμένου Νοεμβρίου και αρχών Δεκεμβρίου πέρυσι και το σχετικό έγγραφο επίσης μας το μοίρασε ο κύριος Χάουαρτ. Περνάμε στον τρίτο μας ο μιλητή κύριο Ράιν Χάρτ από το VCI, την Ένωση Χημικών Βιομηχανιών. Πού είστε κύριε? Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή και για το γεγονός ότι θέσατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη σήμερα, το οποίο με απασχολεί και επαγγελματικά αλλά και ακαδημαϊκά, θα ήθελα σήμερα να θίξω τέσσερα θέματα. Καταρχάς, τα κοινωνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ε, μονομερείς, ε, τα μονομερή μέτρα και σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών στα πλαίσια του ΠΟΕ μέτρα για την τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και θα ήθελα να κλείσω με πέντε συμπεράσματα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Ξέρουμε ότι ο ΠΟΕ και ιδιαίτερα το σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ έχει πλέον αναπτυχθεί και έχει βγει από την κλινική της αυτή φάση και πλέον ισχύουν και άλλοι διεθνείς ε, κανόνες ε, στη διαδικασία αυτή και διαπιστώνουμε ότι πέρα από τις υποχρεωτικές ε, διατάξεις και στον τομέα των περιβαλλοντικών αλλά και στα πλαίσια του ILO η επίλυση των διαφορών δεν υπάρχει με την έννοια αυτή και άρα είναι πολύ ελκυστικός ο ΠΟΕ σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφορών στον τομέα των ε, εμπορικών κανονισμών. Και έχουν καταστεί ιδιαίτερα σημαντικοί αυτοί και ενδιαφέροντες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, έχει οδηγήσει στο ότι ο ΠΟΕ προσανατολίζεται πιο πολύ στα θέματα περιβάλλοντος από ό,τι ισχύει στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου και ο ΠΟΕ στον τομέα του εμπορίου και του περιβάλλοντος λαμβάνει πλέον υπόψη διεθνείς ε, συνιστώσεις. Αυτή η εξέλιξη δεν βλέπουμε να ισχύει για τα εργατικά για τα εργασιακά πρότυπα. Δεν υπάρχουν σχετικέ διαπραγματεύσει στα πλαίσια του ΠΟΑ. Και να θυμίσω στο Υπουργικό Συμβούλιο του 96 στα πλαίσια του ΠΟΕ αποφασίστηκε ότι η αρμόδιος θα είναι μόνος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας, ο ILO. Και η σχετική σύνοδος στο Σιάτλ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο ύψος των προσδοκίων αυτών. Να θυμίσω ότι και το 2001 στα πλαίσια της Ντόχα επαναλήφθηκε αυτό που είχε αποφασιστεί το 1996, δηλαδή η αποκλειστική αρμοδιότητα του ILO. Αν ε, σκεφτούμε τώρα κατά πόσο ο ΠΟΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα, όπως συνέβη και στα πλαίσια του περιβάλλοντος για σε ό,τι αφορά τα θέματα εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων για την ε, τροποποίηση, αν θέλετε, της αντιμετώπιση του ΠΟΕ. Αυτό αποτελεί μια δυνατότητα η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να περάσουν αυτά τα εργασιακά πρότυπα. Το θέμα όμως είναι αν θέλουμε να οριστεί ο ΠΟΕ ως αστυνομία εφαρμογής για τέτοιες συμφωνίες. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τον ILO δεν προβλέπονται τέτοιοι τρόποι επίλυσης διαφορών. Και άρα ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο ο ΠΟΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όργανο ελέγχου. Έχω δύο επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν κατά. Το νομικό επιχείρημα είναι ότι μιλάμε για την ε, διάταξη εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 και κατά πόσον υπάρχει διάσταση εδαφική. Για το περιβάλλον ισχύει αυτή η εδαφική διάσταση, αλλά πιο δύσκολα ισχύει για τις ε, εργασιακά, εργασιακά δικαιώματα. Ωστόσο, θα ήθελα να μην αποκλείσω αυτή τη δυνατότητα στα πλαίσια του ΠΟΕ, αλλά αν χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα στα πλαίσια του ΠΟΕ και τώρα περνάω στο πολιτικό επιχείρημα, θα πρέπει να προωθήσουμε την νομιμοποίηση του ΠΟΕ για να αλλάξουμε την αντιμετώπιση αυτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πολιτική θέληση να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά και σε εθνικό επίπεδο. Και το θέμα είναι αν υπάρχει όντως αυτή η πολιτική θέληση. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι πολιτικά, έχει γενικά κάποιους δισταγμούς και χαίρομαι ιδιαίτερα που η συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί σε εφαρμογή και επεκτείνει τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά θέματα εμπορικής πολιτικής. Γίνονται διάφορες συζήτησεις και κλεισμένων των θυρών. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί το σωστό δρόμο για το μέλλον θα ήθελα να σας πω ότι η μονομερής εφαρμογή σε ό,τι αφορά τα Core Labor Standards στα σύνορα φαίνεται ότι παρουσιάζει προβλήματα. Τώρα, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την τήρηση των ε, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Καταρχάς, ενίσχυση των ε, διεθνών συμφωνιών, κατά δεύτερον διμερείς διαπραγματεύσεις και τέλος ε, θετικά κίνητρα. Τώρα, να περάσουμε στην πολυπλοκότητα των ε, πολυμερών διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι ο ILO θα πρέπει, ε, μάλλον ενισχύθηκε με την δήλωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών στην εργασία του 98, όπου διευκρινίζεται ότι αυτά τα core labor standards θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ακόμα και αν τα κράτη δεν έχουν επικυρώσει όλες τις σχετικές συνθήκες και στην δήλωση κοινωνικής δικαιοσύνης για τον δίκαιο αποκοσμιοποίηση του 2008 διευκρινίζεται ότι ο μη μη τήρηση των προτύπων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα ως προς το κότο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυσικά τα πρότυπα αυτά για προστατευτισμό. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει και το ίδιο σύστημα στον ILO για την επίλυση διαφορών. Δεν υπάρχουν κυρώσεις από στον ΠΟΕ. Στον τομέα τώρα του περιβάλλοντος έχουμε κάποιες συνθήκες και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι η ενδεχόμενη σύγκρουση που προκύπτει μεταξύ μιας συνθήκης περιβαλλοντικής με τον ΠΟΕ επιλύονται πλέον πολύ πιο αποτελεσματικά και δεν ε, παρουσιάζονται πλέον τόσο μεγάλα προβλήματα αλλά και εδώ δεν υπάρχουν συγκρίσιμα μεγέθη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μονομερή μέτρα, θα ήθελα να αναφερθώ στο GSP+, Plus, στο γενικό σύστημα, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, το οποίο ωφελεί 16 χώρες και περιλαμβάνει 6.336 προϊόντα. Και ως τελευταίο μέτρο θα ήθελα να αναφέρω στις διμερείς συμφωνίες και πολλές φορές αναφέρθηκε αυτό ήδη σήμερα να θέσω το παράδειγμα της Κορέας για να διευκρινίσω τι ακριβώς ορίστηκε. Τα μέρη δεν αποσκοπούν την εναρμόνιση των προτύπων τους. Υπάρχει νομοθετική και ρυθμιστική ανεξαρτησία η συμφωνία απόσκοπη στον σεβασμό των ε, κυρίων αυτών εργασιακών δικαιωμάτων και απαιτεί την αποτελεσματική εφαρμογή των συνθήκων του ILO και των διεθνών περιβαλλοντικών ε, συμφωνιών συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφορών υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αν αποκλειστεί αυτή η επίλυση των διαφαρών, επιλέγεται η οδός της διαφάνισης και της συνεργασίας με μια υποχρέωση διαδικαστική και την ορισμό αρμοδίου φορέα για την επίλυση των διαφορών αυτών και σε περίπτωση διαφορών που δεν επιλύονται θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σχετικό πάνελ το οποίο θα υποβάλει μια έκθεση μη δεσμευτική και το αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής είναι μια ήπια πίεση, διαβούλευση και διαφορά, το naming and shaming που σημαίνει δηλαδή ο ορισμός και η δημόσια αποκάλυψη των υπευθύνων. Θα ήθελα να κλείσω με τα πέντε συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή πολιτική τώρα. Καταρχάς, θεωρώ ότι... Ναι, να σας ε, ζητήσω να συντομεύετε, λέει ο Πρόεδρος. Κατά τις διεθνείς ε, συμβάσεις θα πρέπει να τονίσουμε πιο πολύ την επίλυση των διαφορών και την ενίσχυση αυτής στις συμφωνίες αυτές. Δεν θεωρώ, κατά δεύτερον, ότι με την πολιτική απέτησή μας στις διμερείς συμφωνίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ως τώρα ότι ως τώρα έχουν προκληθεί ε, μειονεκτήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η εξέλιξη για το ελεύθερο εμπόριο στην Ασία θα πρέπει, δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί. Τώρα, το κατά πόσον θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις ή κατά πόσο θέλουμε να πετύχουμε τα πρότυπα αυτά με μία ήπια πίεση, θεωρώ ότι παραμένει αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν επιχειρήματα που υποστηρίζουν και τις δύο θέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει την οδό της ήπιας πίεσης για την εφαρμογή των προτύπων αυτών και θεωρώ ότι κατά την επαναδιαπραγμάτευση του, γενικού, του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως ε, τα μονομερή πλεονεκτήματα που δίνονται θεωρούνται δεδομένα και μήπως δεν θα πρέπει στις διμερείς διαπραγματεύσεις να θεωρούνται έτσι δεδομένα. Και τέλος, θεωρώ ότι στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να ορίζονται εμπορικά πρότυπα και αυτά να τη χάνουν διαπραγμάτευση στα πλαίσια του ΠΟΕ. Και μετά να περάσουμε σε θέματα εργασιακά και κοινωνικά και πάλι στα πλαίσια του ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for this extensive... Uh, Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ε, εκτενή παρουσίαση για το παγκόσμιο νομικό προσκήνιο και το νομικό πλαίσιο για τις εργατικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Περνάμε τώρα στη δεύτερη φάση της ακρόασής μας. Θα δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ξεκινώντας από την κυρία Σάιφη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ε, οι παρουσιάσεις τους και πολύ συμπληρωματικές. Θα ήθελα επίσης ε, να υποβάλω μέσα ερωτήσεις. Ε, η πεποίθησή μου είναι ότι από τη στιγμή που θέλουμε αυτή η πρακτική να αλλάξει θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το εμπορικό μας σύστημα και επίσης και ο ΠΟΕ να αναδιοργανωθεί ακριβώς ε, για το περιβάλλον εκεί και το εμπορικό θα πρέπει να είναι ίσο με τα υπόλοιπα δικαιώματα. Θα πρέπει να, να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το σύστημα μεταρρυθμίσεων. Στον κύριο Σαμπαλά θα ήθελα να αποβάλω ένα ερώτημα. Αναφέρθηκε σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό Σιγά σιγά, σταδιακά, αλλά ιδιαίτερα βλέπουμε ότι προχωράει η Κίνα εγκαθίσταται, μπορούμε να το πούμε έτσι, στην Αφρική. Είναι σημαντικό, το διευκρίνησε, είπε ότι για την Κίνα, στην Ήπειρο αυτό, δεν υπήρχαν υποχρεώσεις ε, για τον κύριο Σαμπαλά, μήπως θα μπορούσε να μας εξηγήσει και πάλι πράγματα πάνω σε αυτό και επίσης για τον κύριο Χάουαρντ μια ερώτηση για τις υποχρεώσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μιλήσαμε για παραβιάσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων Επίσης ε, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ε, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι επιχειρήσεις αυτές πραγματικά να σέβονται τις υποχρεώσεις τους και για αυτές τις πολυεθνικές ε, τι θα δημιουργηθεί τις ευρωπαϊκές και οι τρεις επίσης ε, έθιξαν ε, το θέμα των αλλαγών με την συνθήκη της Αβώνας ε, των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Τι θεωρείτε εσείς, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα έπρεπε να υπερασπιστεί σύμφωνα με εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το περιβάλλον και για τα κοινωνικά δικαιώματα στα πλαίσια τα εμπορικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα στον Αρλέμ Δεζίρ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές μας. Θα ήθελα δύο ερωτήσει να τους υποβάλω κυρίως. Να μας πούνε ποια είναι η εκτίμησή τους συγκριτικά αυτές οι ρυθμίσεις ε, που είχαμε μετά από αυτά που είπε το Κογκρέσιο των ΗΠΑ ε, για τις σχέσεις της διμερής ανάμεσα στις ΗΠΑ ε, για περιβάλλον, για κοινωνικά θέματα, το Trade Act όπως αποκαλείται και μας ενδιαφέρει κυρίως για τη συμφωνία με την Κορέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστω και αν ε, λέει ότι αυτές οι ρυθμίσεις για την εφόρα ανάπτυξη της διμερείς ε, συμφωνίες ε, μοιάζουν πάρα πολύ ανάμεσα στους δύο όπως και οι άλλες και για να δούμε πώς θα διαφυλάξουμε τα δικαιώματα και εκεί ανάμεσα στους Αμερικανούς και στις Κορέτες και είναι όμως ακριβέστερα τα σημεία αυτά και θα μπορούσαν να μην ισχύσουν όλα αυτά που έχουν ρυθμιστεί εάν δεν υπάρξουν, αν οι εργατικές αυτές υποχρεώσεις και στα πλαίσια του ΠΟΕ. Εδώ στο ΠΟΕ έχει παγώσει όλη η συζήτηση εδώ και το χρονικό διάστημα από την υπουργική, υπουργική συνάντηση στη Σιγκαπούρη του 1995 και είχε προτείνει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση δικών μας ε, μελών ε, και αυτά που είχαν υιοθετηθεί σχετικά με την εξέλιξη που θα θέλουμε να έχουμε στον ΠΟΕ και στο Εθνές Εμπόριο να συσταθεί μια επιτροπή εργασίας και αξιοπρεπή εργασίας ε, στα πλαίσια των συνεργογείων για το περιβάλλον και που επέτρεψαν ακριβώ να ξεκινήσει, να ξεπαγώσει, θα, να ξεπαγώσει η συζήτηση στον ΠΟΕ εδώ και αρκετά χρόνια και να ε, ισχύσουν αυτά που συμμερίζονται αρκετοί ΠΟΕ για τη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και στο εμπόριο, όλα αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά. Κατά την αποψή σα αποτελεί τη σωστή μέθοδο, συμπληρώνοντα όλα αυτά περί συνεργασία από την Γενική του ΠΟΕ που προχωράει μαζί με το Διεθνέ Γραφείο Εργασία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Είπε ο κύριος Χάουαρντ ε, τις κυρώσεις έδειξε το θέμα αυτό, κάτι που συχνά εξετάζουμε και στα οικονομικά ε, που θα ισχύσουν για αυτές τις κυρώσεις ε, στα όλα πλαίσια της ανάπτυξης αλλά ισχύουν κυρώσεις στα πλαίσια των συμφωνιών με το SPG συν, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Υπήρξε μια κάποια σκέψη τι είδου κυρώσει θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ε, ώστε να εφαρμόζονται πραγματικά, να επιβάλλονται. Είναι βέβαια θέμα πολιτική βούληση. Δεύτερο ερώτημα. Υιοθέτησαν το Trade Act ε, το 2009 με πολιτείε. Έχει καθυστερήσει όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι φρονεί σχετικά με την απόφαση αυτή τη Αμερικανική διοίκηση για το Trade Act. Now it's time listen to... Ο κύριος Higgins τώρα από την ΚΟΕ. Α, κατέφθασε. Thank you, Chairman. Sorry. Um, Ευχαριστώ και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, έχουν ε, φοβερές ικανότητες στο λέγιν και στο να διακηρύσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπόδειγμα δημοκρατίας και ύψης των ε, ηθικών αξιών και όλες αυτές οι ε, αξίες της Ευρώπης θέλουμε να ισχύουν στις εμπορικές μας συναλλαγές και στις διαπραγματεύσεις μας με εταίρους μας που είναι όμως φτωχές χώρες και φτωχές κοινωνίες. Δυστυχώς, Πρόεδρε, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Σε ένα γνωστό ποίημα του T.S. Eliot αναφέρεται ότι μεταξύ της ιδέας και της πραγματικότητας πέφτει μια σκιά. Ε, ο όρτος άνθρωπος ε, ή ο κενός άνθρωπος είναι ο τίτλος του ποίηματος. Και πραγματικά είναι πολύ κενές περιεχομένου όλες αυτές ε, οι αξιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγαλεπίβολες αυτές αυτέ δηλώσεις. Γιατί τελείω διαφορετική είναι η πραγματικότητα του εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και φτωχών χωρών και φτωχών λαών. Η εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών και ε, των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, είναι πολύ διαφορετική η πραγματικότητα. Και οι που έχουμε και από άμεσες επαφές ε, είναι ότι αυτές οι εμπορικές συμφωνίες καταστρέφουν την κοινωνική συνοχή, διαβρώνουν τα κοινωνικά πρότυπα και το περιβάλλον σε πολλές χώρες με τις οποίες ε, έχει συνδιαλλαγές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι χώρες αυτές κατακλείζονται από μαζικής παραγωγής ε, μεταποιημένα προϊόντα και εξοβελίζουν ε, από την ε, τοπική αγορά τους εθνικούς παραγωγούς. Πρόκειται για μια αμυγός εμποροκρατική προσέγγιση. Αν εξετάσουμε τις ε, δραστηριότητες κάποιων πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται, της Ευρωπαϊκή Ένωση που δραστηριοποιούνται στη Λατινική Αμερική και είχαμε κράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και είχαμε και μαρτυρίες κατοίκων από τις χώρες αυτές που υπέστησαν στο πετσί του τις συνέπειες των εγκληματικών δραστηριοτήτων ε, πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη, σε μια φτωχή περιοχή του Βόρειου Περού, μια μεγάλη εξορρυκτική βιομηχανία ε, ευρωπαϊκής προέλευσης ε, καταστρέφει το περιβάλλον, προκαλεί τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές και είναι συνένοχη με το κράτος για την καταστροφή και τη διάβρωση της τοπικής κοινότητας. Ακούσαμε και μαρτυρίες στην ΚΟΕ από τη Βραζιλία για τις καταστροφικές δραστηριότητες μιας ε, σημαντικής πολυεθνικής χαλιβουργίας που έχει έδρα τη Γερμανία και προκαλεί τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές ε, στους αλληλευτικούς πόρους και στο θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή γύρω από το Ρίο Τζανέιρο. Ο δόκτωρ Σάμπαλα παρά είναι ευγενικός όταν μιλά για ένα χάσμα μεταξύ των ε, λόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, συμφωνιών που θέτει επιτάπητο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Εγώ θα έλεγα, θα ήμουν πιο αυστηρό, θα έλεγα ότι είναι υποκρισία, κατάφορη υποκρισία αυτή η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάσταση θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Ο εργαζόμενος πληθυσμός και οι φτωχές μάζες ε, στις χώρες αυτές θα πρέπει να αντισταθούν γιατί στον ε, γενναίο, φαύλο, νεοφιλελεύθερο κόσμο στον οποίο ζούμε η ανταγωνιστικότητα με τους Κινέζους που είναι βάναυσος εκμεταλλευτής ε, του πλούτου και του εργατικού δυναμικού της Αφρικής αν και εμείς συναγωνιστούμε σε αυτά τα χαμηλά στάνταρ την Κίνα, τότε είναι που θα επιδεινωθεί η κατάσταση για τις φτωχές αυτές μάζες. Ενώ θα πρέπει να δώσουμε να ενισχύσουμε αυτές τις μάζες, να αντισταθούν και να ανακτήσουν τον έλεγχο το, του φυσικού τους πλούτου και να μην παίζουμε το παιχνίδι των πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που παραθέσατε το ποίημα του T.S. Eliot. Πολύ χρήσιμη αυτή η μία. Θα ήθελα να δώσουμε χρόνο και στους εμπειρογνώμονες καλεσμένους μας Ας αξιοποιήσουμε την παρουσία τους και τις γνώσεις τους και να περιστούμε σε ερωτήσεις για το θέμα που μας ενδιαφέρει. Ο Κάρλος Σούλτερ από τους Πρασίνους έχει το λόγο. Τώρα σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, Συμφώνησα. Δεν συμφωνώ μαζί σου όταν είπατε στην αρχή οι εμπορικοί μας εταίροι δεν ε, τηρούν ε, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα δικά μας. Αν ε, δούμε τι ΗΠΑ, στη Συμφωνία Ναύτα υπάρχουν τέτοια κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Δεν μου αρέσει η Ναύτα βέβαια, αλλά τουλάχιστον υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ε, σε θέματα περιβαλλοντικής συνεργασίας και στη, στο διοικητική, στη Διοικητική Επιτροπή. Και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούν να αφισβητήσουν εθνικές νομοθετικές διατάξεις που είτε δεν είναι αρκετά αυστηρές είτε δεν εφαρμόζονται σωστά. Και το ίδιο ισχύει και για τα εργατικά πρότυπα. Αν εξετάσετε το παράρτημα της Συμφωνίας ΝΑΦΤΑ, αναφέρεται ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, ελάχιστος μισθός, προστασία των μεταναστών εργαζομένων και το ιδιαίτερα αν έχουμε ε, εμπορικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, τότε εκεί υπάρχει δυνατότητα υποβολής συστάσεων για θέματα ε, πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες ή τα κατάλληλα όρια ρήπανσης, ακόμη και σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η συμφωνία να αυτά προβλέπει πολλούς μηχανισμούς. Οπότε Ήδη ο μείζων εμπορικός μας εταίρος έχει αντίστοιχες ε, ρήτρες στις εμπορικές του συμφωνίες και εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Το Κογκρέσο το 2007 έλαβε μία απόφαση και στο Trade Act των ΗΠΑ αναφέρονται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα ως στο τμήμα εμπορικών συμφωνιών. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να πιστεύουμε ότι θα μας ακολουθήσουν οι ΗΠΑ στις προτάσεις μας αυτές και κάτι τέτοιο θα έχει τεράστια επιρροή στη μεταρρύθμιση παγκόσμιας οργάνωσης εμπορίου. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο και πιστεύουμε ότι ανοίγεται εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Να δράξουμε αυτή την ευκαιρία τώρα και να διευκολύνουμε την ε, λήψη συμφωνίας και για περιβαλλοντικά θέματα. Γιατί αν γίνει παγκοσμίω δεκτή μια τέτοια, θα βοηθήσουμε όλες τις χώρες να υλοποιήσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους του Κιώτο. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Τέλος, ο Πέτερ Σάσνη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Έχω μια απλούστατη ερώτηση για τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες. Πώς βλέπετε τις χώρες της Αφρικής ε, και τις χώρες ΑΚΕ σε ό,τι αφορά την κινέζικη επιρροή, γιατί από τη τίποτα θα αλλάξει θα συνεχιστεί η ανάπτυξη, αυτής της, η ανάπτυξη της Κίνας και η ε, ενίσχυση της παγκόσμιας επιρροής της. Αναφέρθηκε αυτή η μερκαντιλιστική προσέγγιση και φαίνεται πολύ ελκυστική όταν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις που να συνοδεύουν τις συμφωνίες. Αλλά εμείς έχουμε πάρα πολλές δεσμεύσεις ε, και περιορισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει ακόμη να αξιοποιήσει τις εμπορικές της συμφωνίες. Και απέναντι στην Κίνα φαίνεται ότι είμαστε σε δυσμενή θέση. Οτιδήποτε σε θέματα γεωργίας ή ε, πρώτων υλών, οι Κινέζοι τα διαπραγματεύονται πανεύκολα και μάλιστα είναι και πολύ ενδοτική απέναντι σε δικτατορίες, σε αυταρχικούς ηγέτες και σε πολλές φτωχές χώρες. Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα είναι κοινά. Οπότε με, τέτοια, με τέτοιο ανταγωνισμό μάλλον αρνητική εξέλιξη θα έχουμε παρά πρόοδο. Παρακαλώ τους καλεσμένους μας λοιπόν να σχολιάσουν πώς βλέπουν ε, την Αφρική μετά από 20-25 χρόνια από σήμερα. Ωραία, πριν δώσω ξανά το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας, θα ήθελα, για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέσατε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο, την κυρία Γιώργενσεν, τη Γιούλια Γιώργενσεν. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο όμως γιατί χρόνο δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, ευχαριστώ θερμά για τη διοργάνωση αυτή τη δημόσια ακρόαση, που είναι πολύ σημαντική για το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συμπεριλάβουμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και θέματα υφόρου ανάπτυξη στι εμπορικέ μα συμφωνίε. Είναι μαζί μου συνάδελφοι και από τη Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση γιατί έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Οπότε θα ήθελα να ακούσουμε και τους τρεις εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καλύψουμε τις διάφορες πτυχές του θέματος. Έχουμε και εμείς ένα δεκάλεπτο για να κάνουμε τα σχόλιά μας στην ακρόαση. Κατάλαβα καλά. Let's half Όχι, κόψτε κάτι. Το μισό, πέντε λεπτά. Άλλωστε υπήρξε συγκέντρωση της εξουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Να μην αποβεί αυτό εις βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρουσία των συναδέλφων από τις Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Απασχόλησης είναι απόδειξη της αγαστής συνεργασίας που έχουμε μεταξύ των διαφόρων ε, γενικών διευθύνσεων. Η καλεσμένη σήμερα στην ε, δημόσια κρόση μίλησε για πολλά θέματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων και αν έχουμε ένα πεντάλεπτο διατρία, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Οπότε θα περιοριστώ στην προσέγγιση περιβάλλοντος και απασχόλησης στις διμερείς μας εμπορικές ε, συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Εγώ θα αναφερθώ στις εμπορικές πτυχές και οι συνάδελφοι στις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές. Αν είχα περισσότερο χρόνο, πολύ ευχαρίστω να σας ανέφερα πιο διεξοδικέ ε, πληροφορίες. Πάντως, στα πλαίσια της ΔΟΧΑ και της ΠΟΕ έχουμε εντολή και για, περιβάλλον, και για το περιβάλλον. Είναι δύσκολες αυτές οι διαπραγματεύσει, αλλά θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα και σθένος. Στο πλαίσιο του ΠΟΕ, τα θέματα της απασχόλησης ε, διχάζουν τους συνομιλητέ. είναι πολύ ακαθόδη ε, συνεργαζόμαστε και με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Έχουμε επαφές με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ο James Howard αναφέρθηκε στη μελέτη για το εμπόριο, την απασχόληση και το περιβάλλον, που είναι ένα καλό παράδειγμα τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο παγκόσμια διακυβέρνηση για να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων οργανισμών και οργανώσεων. Με αυτέ τι σύντομες λοιπόν παρατηρήσει για το πολυμερές πλαίσιο θα ήθελα να μιλήσω για την προσέγγιση μα στις διμερεί εμπορικέ διαπραγματεύσει. Άλλωστε το θέμα αυτό το έθιξαν και οι Στόχο Στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συμπεριλάβει κεφάλαιο αηφόρο ανάπτυξη και δεσμεύσει για την αηφόρο ανάπτυξη σε όλε τι διμερεί εμπορικέ συμφωνίε που διαπραγματευόμαστε. Και η Κορέα είναι το πρώτο παράδειγμα ενός γενικού κεφαλαίου για τη διαφορά ανάπτυξη. Έχουμε και το Cariform που είναι θέμα οικονομικής βέβαια εταιρικής σχέσης και εκεί έχουμε ευρύτερους στόχους που περιλαμβάνουν και τα αναπτυξιακά θέματα. Αλλά η Κορέα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης μας αυτής. Η συμπερίληψη των κεφαλαίων αυτών σε εμπορικέ συμφωνίε είναι κοινό στόχο με πολλού εμπορικού μα εταίρου και συνεργαζόμαστε με χώρε που εστερνίζονται του στόχου μα προκειμένου να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση και σε... στην ανταλλαγή εμπειριών. Έχουμε στενέ επαφές και με Αμερικανού συναδέλφου αλλά και με Καναδέζους, Ζηλανδού, γιατί και η Νέα Ζηλανδία επιδιώκει παρόμοιου στόχου. Στα κεφάλαια αυτά θέλουμε να επιτύχουμε σαφείς δεσμεύσεις για την τήρηση εργατικών προτύπων, για την αξιοπρεπή εργασία και ο Μάικλ Μόρις από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση θα σας ενημερώσει πιο διεξοδικά. Για το περιβάλλον θέλουμε δεσμεύσεις ε, ως προς τις ε, περιβαλλοντικές συμφωνίες και ο κύριος Λάγκενσδορφ που είναι ε, εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος σα πει κάτι γι' αυτό. Φυσικά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα ρύθμιση τη κάθε χώρα, αλλά έχουμε στόχο να πετύχουμε μια δέσμευση για υψηλό επίπεδο προστασίας που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφέ. και επίση ε, θα θέλαμε να συμφωνήσουμε για αποφυγή ρητρών εξαίρεση και αποφυγή της υποβάθμισης των προδιαγραφών. Ιδιαίτερα με τρόπο που να αντανακλά στο εμπόριο και στι επενδύσει. Υπάρχουν και θέματα συνεργασίας ε, στι εμπορικές μα συμφωνίε και έχουμε ένα τρίτο πυλώνα με βασικές δεσμεύσεις, αρχές και τον τρίτο πυλώνα που είναι το θεσμικό πλαίσιο γιατί αυτό που επιδιώκουμε στα κεφάλαια αυτά είναι να εμπλέξουμε τους εμπορικούς μας εταίρους υπέρ ενός διαλόγου και συνεργασίας με τρόπο που να μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης με τις χώρες αυτές. Και έρχομαι στο θέμα που έδειξαν πολλοί συνάδελφοι. Αν οι κυρώσει είναι η σωστή προσέγγιση ή είναι προτιμότερη μια ήπια πίεση ως πιο αποτελεσματικός τρόπος. Σίγουρα πιστεύω ότι οι κυρώσει δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να υλοποιήσουμε τους ε, αναπτυξιακούς μας στόχους με τους ε, εμπορικούς μας εταίρους. Καταρχήν, ε, ο θεσμικός μηχανισμός ε, που προβλέπει μια εμπορική συμφωνία έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή της. Αν ε, ξεκινάτε διαπραγματεύσεις ε, απειλώντας με κυρώσεις, οι χώρες θα φοβούνται αυτόν τον κίνδυνο κυρώσεων και θα είναι πολύ πιο προσεκτικές. Αν ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις με βάση το διάλογο, με βάση την αναζήτηση ενός κοινού στόχου, με επιδίωξη μιας δέσμευσης από τους εταίρους μας, πιστεύω ότι θα σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο από το να τους απειλούμε με κυρώσεις. Γιατί με την ήπια μέθοδο και οι εταίροι μας βλέπουν ότι είναι προς το συμφέρον τους τέτοιες διαπραγματεύσεις. Και ο στόχος είναι να πετύχουμε τη δέσμευση, όχι να φοβήσουμε τους εταίρους μας. Νομίζω λοιπόν ότι από ουσιαστική άποψη είναι προτιμότερη η ήπια Και αυτό φαίνεται και στη συμφωνία με την Κορέα. Η, η συμφωνία αυτή δεν καλύπτει μόνο θέματα προτύπων Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αλλά και άλλα θέματα από το πρόγραμμα του Γραφείου Εργασίας. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς εφαρμογής, διαπιστώνουμε ότι και στις χώρες που υπάρχει δικαίωμα κυρώσεων, δεν έχει γίνει χρήση αυτού του μηχανισμού σε κανένα τρόπο διακανονισμού των διαφορών μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί κυρώσει. Εμείς στηριζόμαστε στη συνεργασία και τον διάλογο σε εμπορικέ μας συμφωνίε και προσπαθούμε να αναμίξουμε ενεργά και την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω αυτό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της σωστής εφαρμογής. Θέλουμε συνεχή διάλογο. Ναι, προσπαθώ, προσπαθώ να μην μακρηγορήσω. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η ανάμειξη των της κοινωνίας των πολιτών, γιατί για να εξασφαλίσουμε αλλαγές δεν αρκεί η συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Θέλουμε και τον ε, έλεγχο, το δημόσιο έλεγχο, την πίεση που απορρέει από αυτόν, αλλά και τη συμμετοχή των ε, συνδικάτων και βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων έχει στενή συνεργασία, στενή συνεργασία με εκπροσώπους των συνδικάτων των εταίρων μας. Υπάρχει λοιπόν στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί θέλουμε και τον έλεγχο από τους πολίτες που είναι πολύ πιο αποτελεσματικός μακροπρόθεσμα και εξασφαλίζει την υλοποίηση των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης και την τήρηση σημαντικών ε, εργατικών προδιαγραφών. Αυτά ελπίζω να επιτρέψετε και στους συναδέλφους να πούν δύο λόγια. Άντε κανένα δύο λεπτά. Okay ο λόγος του συναδέλφου. Ε, ε, ε, ευχαριστώ, συναδέλφοι. Δύο-τρία σχόλια να κάνω για την γενικότερη αυτή προσέγγιση την οποία υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εργασιακά και για τα FTAs. σε ό,τι αφορά τα, τις τη πολιτική και σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσει των εταίρων μας. Πρόκειται. μία δεσμευτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την οποία όμως έχει ε, ασπαστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχετικό ψήφισμα του 2004. Αυτή η προώθηση της, ε, του κοινωνικού διαλόγου, της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας της ισότητας των φύλων και ξεπερνάει τα όρια των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, των ελάχιστων αυτών εργασιακών δικαιωμάτων. Και γι' αυτό συνάντηκε με το βασικό μας στόχο, το ότι το εμπόριο πρέπει να συμβαδίζει με την βιώσιμη ανάπτυξη. Για θέματα αυτά, λοιπόν, η προσέγγιση των ελεύθερων συναλλαγών περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και άλλων βασικών συνθήκων. Κατά δεύτερον, πέρα από τα πρότυπα αυτά, η επικύρωση και άλλων ε, συνθήκων στα πλαίσια του ILO και κατά τρίτον, σε σύγκριση με άλλες χώρες mm. και την προσέγγιση του ως προς τα FTA, μία δέσμευση για τα πρότυπα αξιπρεπούς εργασίας. Και τα βλέπουμε τα πράγματα και από την άλλη οπτική γωνία. Θεωρούμε ότι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία ότι είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής και τονίζει την συνοχή μεταξύ της κοινωνικής ατζέντα της ευρωπαϊκής πολιτικής και της εμπορικής της πολιτικής. Και επίσης σε πολυμερές επίπεδο υποστηρίζουμε ιδιαίτερα αυτές τις νέες ενδείξεις συνοχής μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΠΟΕ και του ILO. Ένα τελευταίο σχόλιο θα κάνω το οποίο και επιβεβαιώνει αυτά που είπε και η συνάδελφος προηγουμένως εισαγωγικά. Αυτή, αυτό το ευρύ φάσμα αποτελεί ένα επιχείρημα για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή θετικών κινήτρων. Γιατί ξεκινάμε από την πεποίθηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν βασίζεται στην εγχώρια πολιτική ευθύνη στις χώρες εταίρους και θεωρούμε ότι οι μηχανισμοί εποπτείας που περιλαμβάνονται στην προσέγγιση FTA αποτελούν σημαντικό παράγοντα και είναι βασικό η κοινωνία των πολιτών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή εποπτείας. Ευχαριστώ. εγώ Τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους και τις προσκεκλημένες μας. Αρχίζω με τον δόκτορα Σαμπαλά. Σαμπαλά Λα. Ορίστε δόκτορα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ απόλυτα το χρόνο μου. Στο ερώτημα της κυρίας του ΕΛΚ για την Κίνα και την Αφρική. Επαναλαμβάνω αυτά που είχα πει προηγουμένως. Στην Κίνα και την Αφρική συνάπτονται μεταξύ Κίνας και Αφρικής διαφορετικές συμφωνίες από τις συνήθεις. Πρόκειται για συμβόλαια ενοικίασης αγοράς ή μακροχρόνια συμβόλαια που συμπεριλαμβάνουν υποδομές, ε, χρήματα κατευθείαν και άλλα. Επίσης όμως αυτά με όρους ενωσιακούς θα θεωρούνταν ως βοήθεια αλλά είναι καμιά φορά συμφωνίες ανταλλαγής πετρελαίου με ορυκτά ή ανάλογες συμφωνίες με εκείνες που είχε η Γαλλία με τις απικίες της. Οι καθαρά εμπορικές συμφωνίες είναι άλλο πράγμα. Να μην τα συγχαίουμε. Όταν μιλάμε για επιλογή των ε, εταίρων μας. Οι συμφωνίες που συνάπτονται στην Αφρική δεν μπορούν να θεωρηθούν με ενωσιακούς όρους να αναλυθούν. Ούτε για τις αγορές πρώτων υλών. Δεύτερο ερώτημα. Για το χάσμα μεταξύ λόγων και έργων. Είναι νομίζω σημαντικό ότι Οι εμπορικές ρήτρες σε σύγκριση με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές σημειώνουν επίσης μια μεγάλη διαφορά και είναι μονόδρομος. Πρόκειται για αλλαγή των ηθών και συνηθιών της άλλης χώρας αλλά στις ενωσιακές συμφωνίες προβλέπονται υποχρεώσεις και από την πλευρά της Ένωσης. Μεταφορά τεχνολογίας, βοήθεια για τη σύσταση συστημάτων περίθαλψης. Τα αυτά όλα η Ένωση τα έχει διαχωρίσει και τα βάζει σε δέσμες βοήθειας και όχι στις καθαρά εμπορικές συμφωνίες. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις κυρώσεις. Οι οποίες όμως αφορούν το θέμα του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να υποχρεώσουμε τους άλλους να αλλάξουν συμπεριφορά. Και άρα είναι περιορισμένο εύρος, δεν καλύπτουν όλα τα περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά, ούτε είναι αμφίδρομα όλα αυτά όπως ισχύει για τη μεταφορά τεχνολογίας και χορήγηση βοηθείας. Οι κυρώσεις προβλέπουν ότι αν δεν αλλάξουν συμπεριφορά ορισμένες χώρες δεν πρόκειται να υποφεληθούν από την αφίδρομη αυτή σχέση. Ούτε μπορούν οι χώρες αυτές, αν και ορισμένες θα μπορούσαν να επιβάλλουν αντικυρώσεις τα ερωτήματα των κυρίων Δεζήρη και Αρίφη. Η εμπορική πολιτική της Ένωσης στηρίζεται στην εντολή που έχει και καθορίζει απριόρι πριν αρχίσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ότι οι εμπορικές ρήτρες της συμφωνίας, όχι μόνο τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά αλλά τα καθαρά εμπορικά, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές ανάγκες. Αυτό το βλέπουμε και στις οδηγίες για την εργασία και τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Τώρα για τις πολυεθνικές πρώτα. Υπάρχουν δύο πολύ καλά διεθνή εργαλεία, ο ΣΑΚ και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη εφαρμογή, λειτουργία των εργαλείων αυτών. Μέσω παραδείγματο χάρη της συμπερίληψης ρητρών που αναφέρουν οι συμβάσεις των δύο αυτών οργανισμών που έχει συνυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυρώσεις ή άλλοι τρόποι οικονομικής πίεσης γι' αυτά έχουμε να πούμε ότι τέτοιου είδους πιώσεις, πιέσεις έχουν με ένα αποτέλεσμα μέσω της μονομερούς πίεσης που κάνει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων όπως έγινε με τις χώρες του Περσικού κόλπου προηγουμένως ας πούμε που αναγκάστηκαν να αλλάξουν την εργασιακή τους νομοθεσία για να μπορέσουν να διαπραγματευτούν με την Ένωση. Και χώρες όπως το Σαλβαδόρ και η Γεωργία έχουν αποδείξει ότι άρχισαν να σέβονται την εργασιακή νομοθεσία που ισχύει διεθνώς. Διότι είχαν διαγραφεί από τον κατάλογο των χωρών του συστήματος Γενικεμένων προτιμήσεων και για να ξαναμπούν αναγκάστηκαν να επιφέρουν αυτές τις βελτιώσεις. Μπορούν λοιπόν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τις κυρώσεις έμεσες και άμεσες. Και πρέπει τέτοια μέτρα να εφαρμόζονται όποτε χρειάζεται. Ως τελευταία βέβαια, ως τελευταίος έσχατος τρόπος άσκησης πολιτικής, αλλά είναι σημαντικός. Τώρα τα ερωτήματα των κυρίων Ναρίφ και Ντεζίρ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η και ο Καναδάς συμπεριέλαβαν στις διημερείς του συμφωνίες με το Περού και την Κορέα το θέμα προστήμων σε περίπτωση παραβίασης των εργασιακών προτύπων. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Πρώτη φορά προβλέπεται σε τέτοιου είδους εμπορική συμφωνία. Βέβαια για τα πρόστιμα αυτά προβλέπεται να ανακυκλωθούν σε μέτρα μεταρρύθμισης στις χώρες που θα έχουν υποστεί το πρόστιμο και όχι δεν πληρώνονται από τις χώρες που το επέβαλαν, που το ζήτησαν. Πρέπει και η Ένωση να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο, ώστε να συνηθίσουν και οι τρίτες χώρες να συζητούν και να συμπεριλαμβάνουν τέτοια θέματα στις εμπορικές συμφωνίες. Τέλος, το τελευταίο ερώτημα. Η Κίνα και άλλες χώρες που δεν σέβονται την διεθνή εργασιακή νομοθεσία είναι πρόβλημα αλλά μπορούν να ληφθούν μέτρα και κατά αυτόν. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, όχι ίσως πλήρης κυρώσεις, αλλά υπάρχουν άλλα πιο έμεσα μέτρα πίεσης και από τον ΠΟΕ και από αλλού. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον καθηγητή Κουίκ, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και ένα έγγραφο στα γερμανικά που μας έχει υποβάλει και ίσως να ζητήσουμε να μας δώσει και την παρουσίαση του τύπου PowerPoint. Πρόεδρε, θα απαντήσω σε τρία από τα ερωτήματα. Το ένα ήταν η δημιουργία της Επιτροπής του ΠΟΕ για την προετοιμασία των εμπορικών συμφωνιών. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια τέτοια επιτροπή γιατί η υπάρχουσα επιτροπή περιβάλλοντος και εμπορίου έχει βελτιώσει τα πράγματα αλλά εμένα με έχει απογοητεύσει διότι το 96 γράφτηκε μια πολύ καλή έκθεση αλλά από τότε οι υπόλοιπες ήταν πολύ πτωχότερες. γίνονται διαπραγματεύσεις που συνδέουν το εμπόριο με, την, με το περιβάλλον στον ΠΟΕ αλλά δεν καταλήγουν πουθενά μέχρι στιγμής και δεν είναι και δεσμευτικές οι δηλώσεις που γίνονται. λόγω δε του ασαφούς αποτελέσματος του γύρου της Δόχας δεν μπορούμε να έχουμε καμία εγγύηση. Πρέπει στις διμερείς συμφωνίες να υπάρχει μια υποχρεωτική δεσμευτική ρήτρα σεβασμού των περιβαλλοντορικών και εργασιακών προτύπων. Και στις διαπραγματεύσεις που κάνει η Ένωση με πολλούς άλλους εταίρους της θα έπρεπε να ζητάει το σεβασμό αυτών των προτύπων και μόνο σε αυτή την περίπτωση να αρχίζουν διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ. οι διμερείς συμφωνίες δηλαδή να έχουν ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή φυσικά μιας διαφανούς διαδικασίας συνεργασίας και δηλαδή. Να πούμε δηλαδή ρητά στους εταίρους μας ότι θέλουμε να αφισβητήσουμε τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα εφόσον και αν δεν σέβονται τα διεθνή πρότυπα. Από την διμερικότητα καλό θα ήταν να περάσουμε στην πολυμερικότητα. Γιατί μόνο έτσι νομίζω ότι θα μπορούμε, θα είμαστε σε θέση να σταματάμε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αν υπάρχει παραβίαση. Ναι, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από αυτό. Για τις κυρώσεις στις διμερείς συμφωνίες το θέμα είναι τι κυρώσεις προβλέπονται σε μια συμφωνία ε, γενικά ελεύθερου εμπορίου τα ισχύοντα από την Ένωση προβλέπουν την εφαρμογή δασμών ύψους 4% για μένα αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τα δε πρόστιμα δεν νομίζω ότι είναι σωστή ιδέα. Διότι η εναλλακτική λύση δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν λειτουργεί. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερη. Και αφού πάρουμε τα πρόστιμα, τι θα τα κάνουμε τα χρήματα. Τι θα τα κάνουμε. Τέλος το ερώτημα του κ. Στάσνη. Έχω πει και πριν, δεν έχει αποδειχτεί αρνητικό αλλά σκεφτόμουν την Αφρική ας φανταστούμε συμφωνίες μεταξύ ασιατικών χωρών όπου δεν υπάρχει σεβασμός των εργασιακών και περιβαλλοντολογικών προτύπων. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί μια χώρα με την οποία εμείς διαπραγματευόμαστε συμφωνία ελεύθερων εμπορίου την απορρίπτει διότι εμείς επιμένουμε στα εργασιακά και περιβαλλοντολογικά. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα της Ευρώπης. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ χρήσιμη και σκόπιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και συγκεντρώνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για να διαμορφώσουμε πιο εμπεριστατωμένη γνώμη. Ευχαριστώ θερμά τους ε, εμπειρογνώμονές μας που μας αφιέρωσαν τόσο χρόνο στη δημόσια κρόση και σας ευχαριστώ θερμά που μοιραστήκατε τις γνώσεις μαζί μας. Σας διαβεβαιώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για μια σωστή ενημέρωση και περιμένει από τους εμπειρογνώμονες τεκμηριωμένες πληροφορίες για να μπορέσει να συγκεντρώσει απαραίτητα στοιχεία και να συντάσει τις εκθέσεις του. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στην ακρόαση και για τη συμβολή τους στο να γίνει αυτή πραγματικά επικοδομητική και ενδιαφέρουσα. Και εδώ κυρίσω το πέρα στις δημόσιες ακρόσεις, αλλά χωρίς διακοπή θα περάσουμε στην ε, επόμενη, στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 7, θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες, ναι. τροποποίηση του κανονισμού του 1934-2006. Η νομική βάση του, α, της πρώτης αυτής έχει επίσημα τροποποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την ανακοίνωση Omnibus όπως είναι γνωστή και η νέα νομική βάση του αναθεωρημένου κανονισμού είναι ένα συνδυασμός του άρθρου 207 και του άρθρου 209 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα με χαρά να σας ενημερώσω ότι ε, καταλήξαμε σε συμφωνία με την ΑΦΕΤ ε, που θα συνεργαστεί μαζί μας για τα, θέματα αυτά, ε, για τα θέματα αυτά. Στις 26 Ιανουαρίου θα εξετάσει τη γνωμοδότηση η ΑΦΕΤ. Στις 27 θα εξετάσουμε εμείς την έκθεση στην Επιτροπή Διεθνού εμπορίου. 23 Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί στην ΑΦΕΤ. 16 και 17 ε, Μαρτίου θα εγκριθεί έκθεση εδώ. Και 24-25 Μαρτίου ή 9 ε, ή 10 Απριλίου θα περάσει η έκθεση στην Ολομέλεια. Στα τέλη του περσινού έτους και η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ζήτησε να γίνει συνδεδεμένη επιτροπή για το θέμα αυτό με βάση το άρθρο 50 της διαδικασίας. Εγώ απαντώντας στο αίτημα της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, απέριψα το αίτημα στηριζόμενο σε τρεις λόγους. Σε αντίθεση με τους χειρισμούς της ΔΕΒΕ, η τροποποίηση της νομικής βάσης δεν δικαιολογεί την ε, απόδοση του καθεστώτος της Εδεμένης Επιτροπής και στην Επιτροπή ΔΕΒΕ. Γιατί η αλλαγή της νομικής βάσης έγινε αμυγός για τεχνικούς λόγους. Καμία ουσιαστική τροποποίηση δεν έγινε στην αρχική πρόταση. Δεύτερον, και μελλοντική χρηματοδότηση του ICI δεν είναι βάσιμο επιχείρημα για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων. Άλλωστε, ένα σημαντικό τμήμα της χρηματοδότησης προέρχεται από ανακατανομή των κονδυλίων του ΙΣΙΑΙ του χρηματοδοτικού μέσου, κάτι που δεν δικαιολογεί το να γίνει η DEVEP και πάλι συνδεδεμένη επιτροπή για το θέμα αυτό. Άλλωστε, η χορήγηση ενός τέτοιου καθεστώτος στην DEVE θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες διαδικαστικές και πρακτικές δυσκολίες για τη διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, απέριψε το αίτημα της ΔΕΒΕ να συνδεδεμένη επιτροπή. Από ό,τι ξέρω και επειδή δεν έχουμε και πολύ πίεση χρόνου για το θέμα αυτό και απουσιάζουν οι περισσότεροι συντονιστές, θα σας πρότεινα να διαβιβάσω τα σχετικά έγγραφα στους τονιστές μετά το πέρας της συνεδρίασης για να μου πούν τη γνώμη τους. Και να μπορέσουν να μου απαντήσουν το συντομότερο δυνατό. Εκτός φυσικά και αν υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την πρόταση που σας έκανα. Υπάρχουν σχόλια. Ο κύριο Σούλτ καταρχήν. Ο, ο κύριος που είναι και ο εισηγητής ε, για το θέμα αυτό. Ε, Mr. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που αναλάβατε τον τελευταίο μήνα γιατί με την έκθεση αυτή έχουμε πραγματικά μία άνευ προηγουμένου κατάσταση και έστειλε και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ίντα το πρωί το καθεστώς που ισχύει για την επεξεργασία αυτής της έκθεσης. Δηλαδή, σας έστειλε πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο, για την προγραμματισμένη κοινή προσέγγιση στον τριμερή διάλογο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επίσημα έγγραφα που μας έστειλε προς το περιεχόμενο και τα προτινόμενα κονδύλια για το χρηματοδοτικό αυτό μέσο. Συμφωνώ με την προσέγγισή σας, δηλαδή να προσπαθήσουμε αυτή την κατεύθυνση να ακολουθήσουμε και επίσης ε, θα ήθελα να μάθω την άποψη των μελών της Επιτροπής ΙΝΤΑ συμφωνείτε με την πρόταση κάποιος από την Επιτροπή μας να συμμετέχει και να αναλάβει την εντολή να μας εκπροσωπήσει στον τριμερή διάλογο. Καλά, αλλά αυτό το συζητήσουμε στην επόμενη μας συνεδρίαση, γιατί σήμερα δεν έχουμε μεγάλη παρουσία ώστε έχουμε πραγματικά επικοδομητική συζήτηση. Ο κύριος Καντέρ Αρίφ. Πρόεδρε, όχι. για τα λόγια σας ε, γιατί μας ε, είπε ότι ο εισηγητής ε, με την πρόταση για τη μέθοδο από την οποία υποβάλλετε εσείς με την Επιτροπή Ανάπτυξης έγινε μια επαφή και ο, αντι, αντίστοιχος μου εκεί είπε τα κύρια που θα πρέπει να διέπουν τη συμφωνία μας και την σχέση μας ε, για τα θέματα του προπολογισμού. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε αυτά τα χρήματα που θα πήγαιναν ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία με χώρες που δεν χρειάζονται παρόμοια ενίσχυση και από τους φίλους μας της Επιτροπής Ανάπτυξης λένε ότι ηθικά, οικονομικά δεν είναι αυτό απαράδεκτο τα χρήματα που πηγαίνουν για τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης μετά να χρησιμεύσουν για τη συνεργασία με τις χώρες από τις πλουσιότερες ήδη του πλανήτη μας. Δεν είναι ότι διαφωνώ με την πρότασή σας, αλλά από πολιτικής πλευράς, ε, γιατί την εμπορική ανάπτυξη την υπερασπίζουμε όταν όμως είναι θετική και εδώ όλα αυτά που προτείνουμε στον εισηγητή και στον σκιώδη εισηγητή το θέμα αυτό θα πρέπει να εγγραφεί στα πλαίσια απόλυτα των προτεραιοτήτων ο τρόπος τουλάχιστον με τον οποίο θα εκφραστεί η Επιτροπή μας για το θέμα αυτό, για το εργαλείο αυτό δεν ε, θα ακριβώσει περισσότερο, δεν θα εξετάσω περισσότερε λεπτομέρειε, αλλά νομίζω ότι αξίζει περισσότερο από μια τεχνική αντιμετώπιση πάνω σε αυτό το εργαλείο. Στάσνη από το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε. Να δηλώσω τη θέση μας ως ε, ΕΛΚ. Συμφωνούμε με την πρόταση και την πρόταση του εισηγητή. Αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε και μετά να έχουμε και το χρόνο τον απαραίτητο για να το συζητήσουμε και με τους συντονιστές. Ε, Helmut Schultz. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να προσθέσω ένα σχόλιο. Φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε το περιεχόμενο, αλλά το είπα και εξ αρχής ότι από πολιτική άποψη συμφωνώ με τις παρατηρήσεις οι οποίες μόλις έγιναν από τον συνάδελφο Αρίφ θα πρέπει να επιμείνουμε για να συμμετάσχουμε στην διαδικασία λήψη αποφάσεων προκειμένου να μην αφαιρεθούν τα χρήματα αυτά από την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο τριετές. Στην επόμενη περίοδο θα υπάρχει μια νέα προσέγγιση για την αδιάρθρωση των, μεσών, των μέσων. που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να δούμε όλο το πλαίσιο δηλαδή και μετά να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε τη δική μας προσέγγιση. αλλά στην παρούσα φάση να επιβεβαιώσουμε την πολιτική μας δέσμευση και πολιτική μας πρόθεση μαζί με την ε, φυσικά κατανοητή επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει το μέσο αυτό, γιατί, όπως είπατε και εσείς, το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πυκνό τον Ιανουάριο και θα είναι δύσκολο να τηρηθεί το πρόγραμμα, το οποίο φυσικά θα ωφελήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τριτές χώρες. Ο κύριος Καζάκ. Ναι, πρόεδρε θα συμφωνήσουμε και εμείς με την πρόταση την οποία αναφέρατε και του εισηγητού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Γι' αυτό το εργαλείο βέβαια εκφράντως την ευαισθησία μας σε αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν από λίγο. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση γι' αυτό αν υπάρχει συμφωνία, μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση του κυρίου Αρίφ. Αμέσως μετά τη συνεδρίαση πάντως, θα σας μοιράσω τη θέση μου για να καταλάβετε και εσείς καλύτερα το πρόβλημα και για ποιους ακριβώς λόγους ε, επέμεινα στην ε, θέση μου. Συμφωνείτε? Ωραία. Now we move to point Να περάσουμε στο 8 τώρα τη ημερήσιας διάταξη. μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία. Όπως θα θυμάστε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησαν μάλλον διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά ξεκίνησαν ευρύτερες διαβουλεύσει. Ωστόσο, όταν κατέστη σαφές ότι θα δεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνα. στις 23 Νοεμβρίου του περσινού έτου, στην Ολομέλεια, τέθηκε ο όρος η συνθήκη της Λισαβόνα και παραθέτω να, να αποτελέσει την νομοθετική βάση για την μακροοικονομική βοήθεια. Τέλος παράθεσης. Και συγκεκριμένα παράθεσης από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί πλαίσιο νομοθετικό θα γίνουν προτάσεις ε, μακροοικονομικής βοήθειας σε συνεργασία και σε συναπόφαση με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω για την πρόταση αυτή το εξή χρονοδιάγραμμα 27 Ιανουαρίου να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης 16 και 17 Μαρτίου να γίνει ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης και 24-25 Μαρτίου και 2 Απριλίου να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ωστόσο, υπάρχει ένα διαδικαστικό ζήτημα που ανακύπτει αναφορικά με την πρόταση αυτή. Έκανα το σχέδιο έκθεσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχα αναλάβει τότε, αλλά δεν ε, το δημοσίευσα, δεν σας το έδωσα γιατί ανέκυψαν νέες εξελίξεις. Η νομική βάση για την πρόταση αυτή θα έπρεπε να είχε ήδη τροποποιηθεί από την επωνομαζόμενη ανακοίνωση Omnibus παρά τα σχόλια που αποστήλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έγκριση της ανακοίνωσης αυτής, η μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία δεν συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα που χρειάζεται για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκαν, αλλά στο παράρτημα 4 που αποτελεί τον ενδεικτικό κατάλογο της μελλοντικής ε, μακροοικονομικής βοήθειας. Άρα δεν υπάρχει βεβαιότητα για το κατά πόσο το Κοινοβούλιο έχει λάβει την απαραίτητη εντολή για την προετοιμασία της έκθεσης και την ψήφιση της στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν ενώ έχω καταρτήσει την έκθεση δεν την έχω αποστείλει για μετάφραση ούτε την έχω διαβιβάσει στα μέλη της, Ευρω... της Επιτροπής. Και επειδή η βοήθεια αυτή είναι μάλλον κατεπήγοντος χαρακτήρα, θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια σαφή απάντηση. Να μας πει ποια είναι η θέση της για την τρέχουσα κατάσταση και τι θα κάνουμε στο μέλλον προκειμένου να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Για να δω, για να, γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Λουκάστα Μητσιώτη ή στον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο για να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω ποιο από τους δύο θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε επίσης που βάλατε το θέμα αυτό στην ατζέντα. Θεωρούμε ότι είναι καταπήγον το θέμα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επ' ευκαιρία και για την εξαιρετική μας συνεργασία τον ε, περσινό Νοέμβριο. Κινήθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις τέσσερις αυτές προτάσεις που υποβάλαμε ήδη πέρσι. Και φυσικά ελπίζουμε και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Τώρα, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία, για την μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κομισιόν ε, ενέκρινε την πρόταση αυτή στις 29 Οκτωβρίου. Φυσικά από την 1η Δεκεμβρίου έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για ένα νομοθετικό διαδικαστικό θέμα και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή επί της ουσίας της πρότασης. Η κατάσταση παραμένει ως είχε είναι δύσκολη η κατάσταση. Η Ουκρανία χρειάζονται τα χρήματα αυτά. Δεν έχουμε αλλάξει λοιπόν γνώμη και επιμένουμε στην ίδια προσέγγιση. Αυτό είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Okay. You hear me? Με ακούτε τώρα? Μάλιστα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι θα επιμείνουμε στην πρόταση. Εμένουμε στην πρότασή μας, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Δεν έχουμε αλλάξει γνώμη για τα θέματα τα διδικαστικά και τα νομικά σε ό,τι αφορά τη μετάφραση στη νομική γλώσσα της Νέας Συνθήκης. Να πούμε δηλαδή διαμόρφωση της πρότασης στα πλαίσια της Λισαβόνας. Να σας πω σήμερα ότι η πρόταση μακροοικονομικής βοήθειας για την Ουκρανία αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης Omnibus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή θα αποτελέσει τμήμα της απόφασης της ανακοίνωσης αυτής γιατί θα εγκριθεί σύντομα η ανακοίνωση αυτή. Τώρα, για την αλλαγή που θα χρειαστεί στην ανακοίνωση, όντω έγινε ένα πρακτικό λάθος και τοποθετήθηκε το θέμα αυτό στον παρά... στο παράδειγμα 4, το οποίο θα σημαίνει μεγαλύτερη καθυστέρηση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και σήμερα πρέπει να σας ε, διαβεβαιώσω ότι θα μπει στο παράρτημα 1 το οποίο σημαίνει άμεση εφαρμογή της δράσης μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν καθυστερήσεις, χαίρομαι να σας ανακοινώσω σήμερα. Επίσης να σας πω ότι η νομική βάση για τη νέα αυτή πρόταση θα είναι το άρθρο 2.12, το οποίο συνάδει και με τις συζητήσεις που έγιναν και με τις συμφωνίες μας. Άρα από την άποψη αυτή θα χαρούμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας και το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται, το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. για να εγκριθεί η πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ καλές ειδήσει διευκρινίστηκε το πρόβλημα. Άρα θα συνεχίσω τα καθήκοντά μου ως εισηγητής και θα διαβιβάσω αυτή αμέσω μετά τη συνεδρίαση την έκθεση, το σχέδιο έκθεση στα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Ρίγκλερ από το ΕΛΚ. Σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ συντομός. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο στοιχεία. Καταρχάς, εξ ονόματος της ομάδας μας, της Επιτροπής ΙΝΤΑ, ε, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι υποστηρίζουμε το χρονοδιάγραμμα που προτείνετε και όλες τις υπόλοιπες προτάσεις που κάνατε εισαγωγικά στο θέμα αυτό και επίσης σας ευχαριστώ για τις διαδικαστικές πληροφορίες, τις πληροφορίες επί τις διαδικασίες που λάβαμε έξω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι χρειάζεται και μία σύντομη πολιτική δήλωση, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μας υποστηρίζουν το κατεπήγον της πρότασης αυτής, γιατί ουσιαστικά αποτελεί τμήμα των προσπάθειών που κατεβάλλει η Ουκρανία προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Άλλος ε, εκπρόσωπος των άλλων πολιτικών ομάδων θέλει να πάρει το λόγο. Συμφωνείτε λοιπόν για το χρονοδιάγραμμα το οποίο πρότεινα. το οποίο συμφωνήθηκε και στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο των φιλελευθέρων. Μάρτιν Κάζακ, θες να πάρεις το λόγο. Oui, Πρόεδρε, ναι. Επιθυμώ να λάβω το λόγο για το θέμα αυτό το οποίο αναφέρεται και υπάρχουν δυσκολίες για την αντιμετωπίση της πρότασης της Επιτροπής η οποία υπευλήθη για αυτά τα μακροοικονομικά αλλά αναμένοντας την απάντηση του εκπροσώπου της Επιτροπής ικανοποιήθηκα όπως και εσείς από την επίδειξη καλής διάθεσης της Επιτροπής να ενεργήσει, να δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια της ισχύ, της νέας συνθήκης και τη νέα διαδικασία που εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή επιθυμούμε να εφαρμοστεί και αυτό στα πλαίσια αυτών των σχέσεων και αυτής της συμφωνίας. Στον εκπρόσωπο της Επιτροπής να ρωτήσω το εξής. Στη συνάντηση του Κοινοβουλίου της 23 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια ε, μας είχε υποσχεθεί η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την νομοθετική αυτή τακτική διαδικασία ανάλογα με την περίπτωση σε κάθε θέμα που έχει να κάνει με αυτή την αρρωγή τη μακροοικονομική και να περιμένει μέχρι τη στιγμή που θα είχαμε ένα κανονισμό πλαίσιο που θα ρύθμιζε την όλη κατάσταση και θα είχε υιοθετηθεί Υπάρχει ήδη ένα παρόμοιο σχέδιο παρόμοιου ρυθμιστικού πλαισίου και εσείς σαν Επιτροπή πότε προτίθεστε να υποβάλλετε πρόταση παρόμοιου κανονισμού για την Επιτροπή είναι αυτή η ερώτηση. Μήπως, Μήπως υπάρχει κάποια τέτοια πρόταση για το σχέδιο κανονισμού για τα... τη μακροοικονομική βοήθεια. Ευχαριστώ. Όπως είπα και στην τελευταία συνεδρίαση, πρόκειται για ένα σχέδιο που όμως δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε σήμερα, γιατί δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Επιτροπή. Οπότε σήμερα δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τίποτα. Θα επανέλθουμε για το ίδιο θέμα. Θα πρέπει πρώτα να σχηματιστεί η Επιτροπή και να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της. Ε, ναι, είναι εύλογο αυτό το επιχείρημα. Άλλα σχόλια για το θέμα αυτό. Ο κύριος Σόλτς, παρακαλώ, χρόνο φίδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα μικρό, μια μικρή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκλογές ε, στην Ουκρανία δεν αναφέρθηκαν που είναι επικείμενες. Θεωρείτε ότι οι εκλογές αυτές θα αλλάξουν κάτι σε ό,τι αφορά το πλαίσιο αυτό στο οποίο εργαζόμαστε. To the commission, I understand. Το ερώτημα είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν έχει σχόλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της ερώτησης αυτής σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των επικείμενων εκλογών στην Ουκρανία. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά, ασφαλώς. Είναι σαφές ότι οι εκλογές οι οποίες θα διοργανωθούν σύντομα στην Ουκρανία ε, μας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε πριν από τις εκλογές. Έχουμε ήδη ένα μνημόνιο συμφωνίας με την Ουκρανία με τους όρους μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πριν τις εκλογές. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι το χρονικό πλαίσιο δεν είναι ασύμβατο σε ό,τι αφορά δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών και τις συζητήσεις μας εδώ. Νομίζω ότι την άνοιξη ε, εγκαίρως θα μπορέσουμε να προεδράσουμε στο επόμενο βήμα. Μάλιστα, λοιπόν, το σχέδιο έκθεσης μου, λέει ο Πρόεδρος, θα σας διαβιβαστεί αμέσως μετά την συνεδρίαση και θα το συζητήσουμε στις 27 Ιανουαρίου. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 9 για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Σε ό,τι... Συγγνώμη, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν σε ό,τι αφορά τη Σρι Λάγκα. Το οποίο συμφωνήθηκε πριν από αρκετές εβδομάδες. Έχουμε ένα κατάλογο ομιλητών προσκεκλημένων Θα είμαι πολύ αυστηρός γιατί έχω... ...17 λεπτά. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο ευθύς αμέσως στους ε, βασικούς ομιλητές. Δύο ομιλητές για 10 λεπτά. Αλλά θα περικόψω... θα κλείσω το μικρόφωνο μετά από 10 λεπτά και μετά 5-6 λεπτά για τους υπόλοιπους ε, συμμετέχοντες. να σας κάνω κάποια σχόλια για να καταλάβετε ποιο είναι και το υπόβαθρο. Στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων δίνονται προνόμια σε αναπτυσσόμενες χώρες από το 1971 και σε διάφορα το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ δίνονται επιπλέον τελωνιακά προνόμια σε ό,τι αφορά τους ε, σχετικούς δασμούς και σε ό,τι αφορά χώρες οι οποίες εφαρμόζουν ε, αναπτυσσόμενες χώρες που εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα σε ό,τι αφορά την καλή διακυβέρνηση, τα εργασιακά δικαιώματα και το καθεξής. Οι χώρες θα πρέπει να πληρούν φυσικά ορισμένους όρους οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής, να έχουν επικυρώσει και να έχουν εφαρμόσει όλες τις ε, διατάξεις στο παράρτημα 3, να έχουν επικυρώσει και εφαρμόσει τις σχετικές συνθήκες και να έχουν εφαρμόσει την νομοθεσία και τα μέτρα τα εργασιακά και τέλος να θεωρούνται χώρα ευάλωτη και προβλέπεται η προσωρινή απόσταση, αναστολή των προτιμήσεων αν δεν τηρούνται οι όροι αυτοί ή αν η νομοθεσία δεν εφαρμόζονται επαρκώς. Η Σρι Λάγκα τώρα έχει ωφεληθεί από το GSP+, Plus, από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, από το 2005 και μετά υπό το φως των ε, στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι υπήρχαν ε, λόγοι να ξεκινήσουν έρευνες για τα, την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα το 2008. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η σχετική ε, έρευνα και στις 19 Οκτωβρίου του 2008 υποβλήθηκε η σχετική έκθεση. Η εθνική λοιπόν κυβέρνηση της Σρι σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμβάσεις, ιδιαίτερα για παράδειγμα την συνθήκη κατά των βασανιστήριων και τη συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν τηρούνται λοιπόν όλες αυτές οι συνθήκες στην Σρι Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε λοιπόν μια πρόταση για την προσωρινή αναστολή των ε, επιπρόσθετων προτιμήσεων προς τη Σρι και τώρα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να εγκρίνουν την πρόταση αυτή. Αν εγκριθεί η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ισχύσει μετά από έξι μήνες, όπως προβλέπεται στο σύστημα γενικών, γενικευμένων προτιμήσεων. Θα υπάρξει συναπόφαση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και ασχολείται ιδιαίτερα με την απόφαση αυτή. Η Επιτροπή μας λοιπόν διοργάνωσε μία ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων με τον ε, πρέσβη της ε, Σρι Λάνκα και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ανυπομονούμε να ακούσουμε λοιπόν τους πολύ εμπειρούς ομιλητές πέρα από τον πρεσβευτή της Σρι Λάνκα. Να καλωσορίσω τον κύριο Αριαζίν, πρέσβη της Σρι Λάνκα. και τον κύριο Χάιζεν, διεθνή εκπρόσωπο της ε, οργάνωσης αλληλεγγύης. Και μετά έχουμε και τον κύριο Γκρέι του Βρετανικού Ομίλου και του κύριου Γκράσελ των ε, δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους δύο κύριους ομιλητές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτή που βρίσκεται εδώ πέρα μαζί μας. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Το πολύ δεκα λεπτά σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Η Σρι Λάνκα χαίρεται για την ευκαιρία αυτή να ακουστεί η φωνή της για αυτό το σημαντικό θέμα μετά από μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο της ιστορίας της λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να ερευνήσει τα συμβαίνοντα στη Σρι Λάγκα αλλά εμείς αρνηθήκαμε μια τέτοια παρέμβαση γιατί τη θεωρήσαμε άχρηστη διότι υπήρχαν ήδη άλλα εργαλεία επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ Σρι Λάγκας και ευρωπαϊκών θεσμών. Γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη του καταλόγου των γενικευμένων προτιμήσεων που έχουν σημειώσει παραβιάσεις σοβαρότερες από εκείνες για τις οποίες κατηγορείται η Σρι Λάγκα. Παρ' όλα αυτά αφού έχει ακουστεί η κατηγορία ότι δεν ανταποκρίνεται η Σρι Λάγκα και δεν σέβεται τα προβλεπόμενα από την Ένωση, θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτό είναι ανακριβές. Συνεχίζουμε επιμελώς να τηρούμε όλα όσα έχουν προβλεφθεί στις σχέσεις μας μέσω των διπλωματικών καναλιών με την Ένωση. Και νομίζουμε ότι σε μια αντικειμενική διαδικασία θα μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουμε ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της Ένωσης. Όσο η έρευνα αυτή έγινε μάλλον σε μια ιδιαίτερα όπως είπα ταραγμένη περίοδο της ιστορίας της Σρι Η κατάσταση όμως από τότε έχει ιδιαίτερα βελτιωθεί διότι ιτήθηκε το κόμμα των τίγρεων του Ταμίλ και όλα αυτά είναι γνωστά και δημοσιευμένα. Η Σρι έδωσε τα σχόλια που ζήτησε για τις εξελίξεις αυτές η Κομισιόν και καθόρισε ότι μετά από ενδελεχή έρευνα η Κομισιόν είχε εφαρμόσει επιλεκτικά και διακριτικά την έρευνα που είχε κάνει σε σύγκριση με άλλες χώρες συγκρίσιμες και μετά από αυτά η βελτίωση της κατάστασης στο θέμα της εσωτερικής έντασης αναγνώρισε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη θετική αυτή εξέλιξη και αυτό δείχνει ότι η Σρι Λάγκα κινείται προς την κατεύθυνση της ελληνικής επίλυσης του, της διαμάχης. έχουν βελτιωθεί τρομερά οι αριθμοί όπως θα δείτε στα έγγραφα αυτά των εκτοπισθέντων από τις 284.000 σε μόλις 8 οι τόποι εγκατάστασής τους έχουν τύχει επισκέψεων και από οργανώσεις και δεν βρήκαν τίποτε να προσάψουν. Οι παιδομαχητές έχουν αφοπλιστεί μόνο ένα παιδί από το Δεκέμβριο 2008 μόνο ένα παιδί έχει αναφερθεί ότι έχει γίνει πολεμιστής των τίγρεων του Ταμούλ. Έχει γίνει και προεδρική έρευνα διαταχθεί για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τελευταία φάση της σύραξης ή διαμάχης και δεν έχουμε μάθει τίποτα για νέες απαγωγές και εξαφανίσεις. Τρει τρεις φορές ακούσαμε ότι συνέβησαν επιθέσεις σε σύγκριση με πολλές δεκάδες τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια και μία μόνο επίθεση είναι κάτι που δεν θα το ανεχθούμε. Η ιστοσελίδα του οργάνωσης των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα από το Σεπτέμβριο του 2009 μόνο μία επίθεση σημείωσε. Και η κυβέρνηση έχει δηλώσει σαφώς ότι η δικαστική διαδικασία θα ακολουθηθεί σύμφωνα με τον νόμο και με δικαίωμα έφεσης. Όπως είδατε ο κύριος της Ενάιγκαμ ε, απελευθερώθηκε μετά από την επιβολή του νομισμένου ποσού. Όλα τα νόμιμα κόμματα στη Σρι Λάνκα συμμετέσχουν ισότιμα στις εκλογές και η ομάδα που λέγεται αλληλεγγύη του Ταμίλ που είναι παρούσα σήμερα εδώ αλλά ζητάει μποϊκοτάζ των εκλογών. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι μειονότητες γίνονται σεβαστές στη Σρι Λάνκα και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που διαδίδει η διασπορά. Όλες τις, οι περισσότερες ανησυχίες που έχουν ακουστεί λοιπόν δεν είναι βάσιμες και θα έπρεπε η Σρι να συμπεριληφθεί εκ νέου στον κατάλογο των χωρών με γενικευμένες προτιμήσεις. Ελπίζαμε η Ένωση να λάβει σοβαρά υπόψη της τις αλλαγές αυτές και να εκτιμήσει δεόντως τα αποτελέσματά τους, δηλαδή τη συμπερίληψη της Σρι Λάγκα στον κατάλογο. Αλλά απογοητευτήκαμε από τη σύσταση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο να μην γίνει η συμπερίληψη αυτή ακόμη. Και τελικά, στα πρόθυρα μάλιστα των τελευταίων εκλογών, η απογοήτευση αυτή μεταφράστηκε και εκλογικά. Η Σρι Λάγκα όμως έχει αποδείξει και τις αξίες που επιβάλλει και έχει σταθερούς και ιστορικούς δεσμούς με την Ένωση ώστε να μπορούν να επιληθούν από κοινού τα προβλήματα με τρόπο που να μην ζημιώνει τα συμφέροντα της Σρι Λάγκας. Εμείς δεν ζητάμε ανεφάρμοστα πράγματα και στόχους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ένωση. Γιατί πολλές φορές τα παράπονα εξυπηρετούν εσωτερικά συμφέροντα και πολιτική. Η αναβολή της συμπερίληψης της Σριλάνκα στο κατάλογο θα δυσκολέψει τα πράγματα στη χώρα και θα ζημιωθούν ιδιαίτερα οι εργαζόμενες γυναίκες. Ιδιαίτερα στους νέους τομείς όπως την πορκελάνη, την αλληλεία κλπ. Δυστυχώς παρά τα όσα λέει η Ένωση για τη θέλησή της να βοηθήσει τη Σρι Λάγκα, μετά την αντιμετώπιση του τσουναμίου ας πούμε, ε, τα πράγματα δεν διευκολύνονται. Ο λαός της Σρι Λάγκα περιμένει ακόμα κύριε Πρόεδρε. Μετά από μια τριακονταετή ε, διαμάχη και τις ζημιές που υπέστημεν από το παλιριακό κύμα δεν θα έπρεπε χωρίς λόγο στην ουσία να, να, να αναβάλλεται και πάλι την συμπερίληψή μας στον κατάλογο. Πρέπει να το δεχτεί αυτό η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτά τα εμπορικά μέτρα είναι απλώς τεχνικά και πρέπει αυθαίρετα να χρησιμοποιούνται σαν πολιτικά όπλα, αλλά να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η επίπτωσή τους και κοινωνικά όχι μόνο οικονομικά. Αφού η Ένωση δείχνει μεγάλη κατανόηση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και άλλων χωρών του καταλόγου των γενικευμένων προτιμήσεων, γιατί δεν το κάνει και για τη Σιρλάνκα. Μερικούς τους βολεύουν, άλλους όχι. Η Σρι Λάνκα όμως διατηρεί τις ελπίδες της ότι τελικά θα υπερισχύσει ο κοινό νους και η λογική. Γιατί έχουμε αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα και σε άλλες περιόδους της ιστορίας μας ιδιαίτερα ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προάσπιση της δημοκρατίας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι λογική η έκκληση που απευθύνουμε εδώ στα μέλη της Επιτροπής μετά και από τη θέση ενισχύει τη συνθήκη της Λισαβόνας να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρήσει το θέμα της συμπερίληψης της Σρι όπως της αξίζει. Σας ευχαριστούμε. Έχετε Είχετε εξαντλήσει το δεκάλεπτο και το ξεπεράσετε κατά πολύ μάλιστα το δεκάλεπτο που σας είχα θέσει. Ας ακούσουμε τώρα το δεύτερο μεσομιλή, τον κύριο Σέναν, που είναι ο διεθνής συντονιστής ε, του κινήματος αλληλεγγύης του Σταμίλ. Έχετε το λόγο και σας θέρμο παρακαλώ 8 με 10 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτέ. Η, η τρέχουσα κατάσταση του Σρι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύγχρονο ολοκαύτωμα. Έχουμε εθνοκάθαρση, δολοφονίες, ε, σφαγές, διώξεις τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι στις τελευταίες μήνες του πολέμου η κυβέρνηση σκότωσε 7.000 μαχοπληθυσμό και πάνω από 100.000 άνθρωποι είναι κρατούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ε, είναι από τις χειρότερες καταστολές ε, και μάλιστα η πρόσβαση στα στρατόπεδα αυτά κράτησης για τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους απαγορεύεται. Μόνο η ε, συνοδευόμενοι δημοσιογράφοι ή δημοσιογράφοι φιλοκυβερνητικοί επιτρέπεται να επισκεφθούν αυτά τα κέντρα και μάλιστα όσοι έχουν απελευθερωθεί μετά από εξάμεινο στα ε, κέντρα αυτά ε, έχουν σημάδια στο σώμα τους που δείχνουν τη χρήση βασανιστήριων. Είχαμε επαφές με ορισμένους κρατούμενους και έχουμε πληροφορίες ότι κανένας δεν επισκέπτεται, παραλαμβάνω, αυτά τα στρατόπεδα κράτησης και σίγουρα όχι οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει καν δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των κρατουμένων, δεν μπορούν να εξιστορήσουν τις αποτρόπες εμπειρίες τους και υπάρχουν κάποια άλλα κέντρα διαμετακόμισης με εξίσου απάνθρωπε συνθήκες με τα κέντρα ε, κράτησης. Επίσης υπάρχει στενή παρακολούθηση από το στρατό και για να έχει κανείς πρόσβαση ε, πρέπει να έχει ειδικέ ε, ταυτότητες, διαφορετικές από τις εθνικές ταυτότητες. Έχουμε ένα ανοιχτών φυλακών για τη μειονότητα του Ταμίλ. Ο Κρίστοφερ Πάτερν, ο πρώην Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις, ε, ε κατήρτισε λεπτομεριακή μελέτη για το θέμα αυτό διαπιστώθηκε ότι πάνω από 13.000 νέοι άνθρωποι ε, κρατούνται σε ειδικά κέντρα και το τι συμβαίνει σε αυτά τα κέντρα δεν αποκαλύπτει από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένα μητρό, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, δεν υπάρχουν καν στοιχεία των κρατουμένων στα κέντρα αυτά. Και ο Υπουργό ε, Τεχνολογίας και Επιστήμης επίσκεψη στο Λονδίνο είπε ότι ακόμη και 8χρονα παιδιά κρατούνται σε αυτά τα κέντρα, στα ε, τόπεδα συγκέντρωσης, στα κέντρα βασανιστήριων. Μάλιστα είδαμε κάποια βίντεο κλιπ με βάναυσες εκτελέσεις και βασανιστήρια κατακρατουμένων. Είχαμε και μια γυναίκα τα Μιλ που δολοφονήθηκε ολόγυμνη. Έχουμε αποτρόπες σκηνέ από τα κέντρα αυτά και όσοι κατάφεραν να διαφύγουν από τα κέντρα ε, μας έδωσαν ανατριχιαστικές μαρτυρίες για βιασμούς, βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση. Υπάρχει μια χαρακτηριστική πολιτική καταστολής και κατάργησης. Είδαμε στο Κολόμπο πρόσφατα κάποιον που τον καταδίωξαν μέχρι που έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Υπάρχει καταστολή και των αντιφρονούντων, της αντιπολίτευσης των δημοσιογράφων κάποιο καταδικάστηκε για 20 χρόνια, ένα δημοσιογράφο, μόνο και μόνο επειδή συνέταξε ένα αντικυβερνητικό άρθρο. Ένα άλλο ακτιβητή δημοσιογράφος ε, που κατήγγειλε την ε, βαναυσότητα της κυβέρνηση, δολοφονήθηκε από φιλοκυβερνητικέ δυνάμεις. Είναι μια τραγωδία αυτή η καταστολή που υφίστανται οι αντιφρονούντες και οι αντικυβερνητικοί. Και μάλιστα ένας ακτιβιστής ε, αρνήθηκε την πρόταση να έρθει στην Επιτροπή σας από φόβο για αντιπερίσπασμο. Εγώ ήρθα επειδή ε, ούτως ή άλλως ζω στην εξορία, αλλά και άλλους να προσκαλούσετε θα φοβούνταν να έρθουν. Ένας άλλος ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας Ταμίλ δήλωσε ότι η πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία είναι η πιο βίαιη στην ιστορία του Σιριλάνκα και έχουν δολοφονηθεί ήδη αρκετοί ακτιβιστές. Και είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι το κίνημα αλληλεγγύη τα μίλη ζητά μποϊκοτάρισμα των εκλογών. Αυτό που λέμε είναι ότι ο υποψήφιος Φονσέκα δεν δίνει καμία εναλλακτική λύση για το λαό τη Σρι Και δεν υπάρχει καμία πρόταση για τη βελτίωση της κατάστασης και του βιωτικού επίπεδου στη Σρι Λάγκα. Η παρούσα κυβέρνηση κάνει κατάχρηση της εξουσίας της προκειμένου να εξασφαλίσει επανεκλογή και νίκη στις εκλογές. Η κυβέρνηση του Σρι Λάγκα υποτίθεται ότι ε, αντιμάχεται την τρομοκρατία. Και η Ταμίλ είναι κατά της τρομοκρατίας και δεν συμφωνούμε με τις μεθόδους των Τίγρεων Ταμίλ. Καταδικάσαμε μάλιστα τις δράσεις των Τίγρεων Ταμίλ Είμαστε υπέρ τη ανάληψη δημοκρατική δράση. Πάντως τίποτα δεν συγκρίνεται με την κρατική τρομοκρατία στην Σριλάνκα και τα πογκρόμ που γίνονται κατά μειον, ε, της μειονότητας στα ΜΙΛ. Το κράτος της Σριλάνκα δεν θα κατάφερνε ε, τη νίκη κατά το Ταμίλ αν δεν είχε τη βοήθεια της Κίνας, της Ινδίας και του Πακιστάν έχει σκοτώσει χιλιάδες αθώους η κυβέρνηση της Σρι Όλες αυτές οι χώρες βοήθησαν την κυβέρνηση της Σρι και λέρωσαν με αίμα τα χέρια τους συμμετέχοντας σε βομβαρδισμούς και σε δολοφονίες. Η κυβέρνηση του Σρι καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και βάλεται κατά των θεμελιωδών ελευθεριών. Είναι τελείως διεφθαρμένη και ικανή για όλα. Γι' αυτό και είναι σωστό να αποσυρθεί το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Η Λάγκα είναι η πιο στρατιωτικοποιημένη χώρα της περιοχής και έχουμε πολυάριθμες εκθέσεις που αποδεικνύουν ότι η Σρι Λάγκα βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου της παραβίας ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το GSPC είναι οποιαδήποτε άλλη βοήθεια προς την κυβέρνηση της Σρι Λάγκα θα βοηθήσει στο διαονισμό αυτών των φρικαλαιοτήτων που διαπράττονται εκεί. Και κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως δεν ωφελεί τα θύματα. Οι εργαζόμενοι στην κλωστοϊφαντουργία που έμειναν άνεργοι μετά το τσουνάμι έμειναν αβοήθητοι. Περιμένουν ακόμη επιδόματα επιβίωσης ή επανεγκατάστασης η κυβέρνηση δεν έκανε καμία σοβαρή προσπάθεια για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους παρά τα κονδύλια που επιδαψίλευσε η Ένωση και τις διάφορες ενισχύσεις που έλαβε. Και μάλιστα ο πρόεδρος που είναι μέλος μιας δυναστείας μαζί με την οικογένειά του ουσιαστικά καταστρατηγεί τα δικαιώματα του, του λαού. Φαίνεται ότι η οικογένεια αυτού του βασιλέα είναι η πλουσιότερη της περιοχής όλες οι ενισχύσεις ε, και οι παραχωρήσεις θα χρησιμοποιηθούν κατά του λαού. Οπότε η απόσυρση του GSP Sin είναι ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, αν και δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να στυλιτευθεί η κυβέρνηση και οποιαδήποτε προσπάθεια βοήθειας προς τη Σρι θα πρέπει να μποϊκοταριστεί. Αν θέλετε να βοηθήσετε το λόγο της Σρι θα πρέπει να δώσετε άμεση ενίσχυση σε αυτούς είτε μέσω των ε, οργανώσεών τους. Όχι μόνο οι μουσουλμάνοι και άλλες κοινότητες ε, έχουν ε, εξοργιστεί με την συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση. Δεν προτείνεται καμία πολιτική λύση από την κυβέρνηση αυτή. Μόνο φρικαλαιότητες διαπράττονται και θα, συνεχίσουν, θα συνεχιστούν και στο μέλλον άσχετα με το ποιος θα νικήσει στις εκλογές. Έχουν κατηγορηθεί υποψήφι των εκλογών για παραβίαση, μαζική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι κατεβαίνουν στις εκλογές. Προσοχή λοιπόν, όταν λάβετε τις αποφάσεις να έχετε υπόψη το λαό του, του Σρι Λάνκα. Γιατί 250.000 άνθρωποι ε, κρατούνται σε κέντρα, σε στρατόπεδα κράτησης η ημιότητα Ταμίλ διώκεται ανελαίητα. Η κυβέρνηση της Σριλάνκα βάλεται κατά του ίδιου του, του, λαού. Αυτά πιστεύω να τα λάβετε υπόψη όταν αποφασίσετε για την παράταση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τις ομιλίες. Είχαμε μάλλον δύο ομιλίες από, τις, από αντίθετες πλευρές, από τις αντιμαχόμενες. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνεδρίασή μας και αν θα ήθελε να λάβει το λόγο. Αν θέλετε κι εσείς να ακουστείτε σε αυτήν την ακρόαση. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομα σχόλιο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για τη συζήτηση αυτή. Αν θέλετε να σχολιάσουμε τώρα Ευχαριστώ. Αν πάλι προτιμάτε να περιμένουμε μέχρι του μιλήσουν και οι άλλοι για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ και πάλι. Οπότε από εσά εξαρτάται. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. να ξεκινήσει η συζήτηση και όπως συμφωνήσαμε και στην προηγούμενη συνάντηση της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής μας έχουμε καλέσει και δύο εξωτερικά μέλη που θα συμμετέχουν στη συζήτηση. Τους δίνω λοιπόν το λόγο για πέντε λεπτά. Ο κύριος Γκρέι καταρχάς, που ο οποίος είναι διευθυντής του Βρετανικού Ομίλου λιανεμπόρων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Βρετανικός Όμιλος ε, Λιανεμπόρων είναι εκπροσωπεί περίπου το 80% της αγοράς στη Βρετανία και κάποια από τα μέλη μας ε, προμηθεύουν τη Σρι Λάνκα εδώ και κάποια χρόνια ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τομέα της κλωστού υφαντουργίας. Θα διαιρέσω την ομιλία μου σε δύο τομείς. Καταρχάς, γιατί αγοράζουμε από τη Σρι Λάγκα και κατά δεύτερον, δύο λόγια για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Η Σρι Λάγκα από παραγωγό κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων έχει μεταλλαχθεί σε αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή ένα παραγωγό με προστιθέμενη αξία. Και βασίζεται στην ε, διαμόρφωση την δεντολογική, αν θέλετε, του εμπορικού της χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και περιβαλλοντικά πρότυπα. Η Σρι Λάγκα και η Ασία γενικότερα αποτελεί ε, μία από τις πιο καθαρές γραμμές παραγωγής. Τώρα σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα και την τήρηση της βιωσιμότητας και των σχετικών κριτηρίων έχει ανοίξει πολλά, πολλές άγορες για τη χώρα και έτσι κατάφερε να διαφοροποιηθεί από άλλους προμηθευτές χαμηλού κόστους. Και αυτό είχε φυσικά και ένα τίμημα για το μέλλον του κλάδου στη Σρι Λάγκα γιατί έχει ανεβάσει το κόστος σημαντικά και τα περιθώρια τα οποία έχουν πολλή παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων στη Σρι Λάγκα είναι πολύ περιορισμένα οποιοδήποτε καταναλωτή και να ρωτήσετε θα σας πούν ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τον απασχολούν ιδιαίτερα, αλλά το θέμα είναι αν είναι διατεθειμένο ο καταναλωτής να τα πληρώσει. Και αυτό ασκεί πίεση στους παραγωγούς της Σρι Λάνκα. Αυτά σας τα λέω για να σας παρουσιάσω το υπόβαθρο και να σας εξηγήσω γιατί είναι τόσο ελκυστική ως χώρα για μας η Σρι Λάγκα τώρα σε ό,τι αφορά την αναστολή του GSP+. Θα πρέπει να δούμε την αλυσίδα παραγωγής με δύο διαφορετικούς τρόπους γιατί ο αντίκτυπος είναι διαφορετικός σε κάθε περίπτωση. Η βασική αλυσίδα παραγωγής και μετά έχουμε την κάθετη αλυσίδα για την ε, γενική αλυσίδα, την οποία χρησιμοποιούν οι πιο πολλοί λιανέμποροι, χαρακτηρίζεται από διάφορα στάδια παραγωγής, διάφορους φορείς που εμπλέκονται και πολύ απλά ο λιανέμπορος αγοράζει ένα έτοιμο προϊόν ένδυσης. και έχει να κάνει με την εξωτερική ανάθεση, την κερδοσκοπική εξωτερική ανάθεση της παραγωγής όπου ο ενδιάμεσος φορέας ψάχνει να βρει τον πιο οικονομικά συμφέρον, συμφέροντα παράγοντα. Και αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με το GSP+. Ναι, φυσικά είναι σημαντική η τιμή, όπως και τα θέματα, τα βιντεολογικά, τα περιβαλλοντικά. Η τιμή αποτελεί το βασικό κίνητρο. Στην συγκεκριμένη λοιπόν αλυσίδα παραγωγής που αποτελεί περίπου το 70% του εμπορίου φαντουργία μεταξύ Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και Σρι Λάγκα. Νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει γιατί θα προωθήσει την παραγωγή και το εμπόριο σε άλλες χώρες όπω το, Βι... Βιετνάμ, την Ινδονησία και τον Μπαγκλαντέ. Τώρα, το κάθετα ενοποιημένο σύστημα παραγωγής το οποίο ανέφερα θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστεί από την αναστολή του GSP+. Πρόκειται για μάρκες οι οποίες έχουν επενδύσει σοβαρά στη Σρι Λάνκα, που είναι δικά τους εργοστάσια ουσιαστικά που παράγουν τα ενδύματα στην Σρι Λάνκα. Άρα αυτοί δεν θα επηρεαστούν. Θα σημαίνει φυσικά κάποιο οικονομικό κόστος για αυτούς, αλλά η εστίαση στην βιωσιμότητα και στα περιβαλλοντικά κριτήρια δεν θα είναι κάτι το οποίο θα τους αποτρέψει τώρα. Εγώ θεωρώ ότι πολλοί από τους πελάτες μου θα χρεοκοπήσουν. Πολλοί έχουν χρεοκοπήσει και πέρσι. Θεωρώ ότι οι καταναλωτές δεν πρόκειται να πληρώσουν το επιπλέον κόστος της βιωσιμότητας. Οι τράπεζες θα, δεν θα τηρήσουν τις συμφωνίες πίστοσής τους και Νομίζω ότι η αναστολή του GSP Plus ως παραγωγός της Sri Lanka θα αποτελούσε επιπρόσθετο παράγοντα πίεσης για τις μελλοντικέ μου εργασίες. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπράσελ από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα για να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για τη Σρι Λάνκα την ίδια, αλλά και για τη σχέση μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της καλύτερης κυβέρνησης και της δημοκρατίας. Όταν ε, ξεκίνησε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλαμε μία έκθεση και τότε, πριν από ένα χρόνο και περισσότερο, η κατάσταση ήταν τραγική. Απαγωγές, ξυλοδαρμοί, λογοκρισία, για τους ε, δημοσιογράφους, για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κυβέρνηση η... τα αριθμητικά στοιχεία ουσιαστικά έχουν βελτιωθεί. Τα πράγματα ήταν χειρότερα πριν από ένα χρόνο. Αλλά δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και ότι έχει εφαρμόσει πραγματικά όλες τις δεσμεύσεις, όλες τις υποσχέσεις που άπτονται θεμάτων της έρευνας αυτής. Ήταν σημαντική για δύο λόγους ε, αυτή η έρευνα. Γιατί, καταρχάς, ακούστηκαν όσα είχαν να πούν όλοι οι ακτιβιστές ε, στη Σρι Λάνκα. και όλα όσα διατείνονταν για μη σεβασμό από την κυβέρνηση των διεθνών συμβάσεων. Ήταν πολύ σημαντική επίσης γιατί άσκησε πίεση. Και νομίζω το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ ο πρέσβης σήμερα για να εξηγήσει τη στάση της κυβέρνησής του αποτελεί ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Αυτό που επιδιώκαμε ήταν η ελευθερία της έκφρασης και τα βασικά δικαιώματα του πολίτη να γίνουν σεβαστά το συντομότερο δυνατόν. Ιδιαίτερα εν ώψη και των επικείμενων εκλογών σε δύο εβδομάδες. Δυστυχώς, καταγράφονται πολλές παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου τους τελευταίους μήνες. Αναφέρεται είπε ο πρέσβης μόνο μία τέτοια περίπτωση στο, στην ιστοσελίδα μας. Κοιτάξτε, επειδή δεν το βγάζουμε στην ιστοσελίδα μας δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν τέτοιες παραβιάσεις. Χτες, χτες μόλις. Έγινε ξυλοδαρμός ε, μίας δημοσιογράφου του BBC από εκπροσώπους ενός ε, υπουργού επειδή κάλυπτε την προεκλογική εκστρατεία και χτες η δυνάμεις ασφαλείας πήγα στο γραφείο ενός ε, ηγέτη, ενός διευθυντή μιας εφημερίδας που καλύπτει το ιστορικό υπόβαθρο της χώρας και μάλιστα ο προηγούμενος διευθυντής ε, δολοφονήθηκε πριν από ένα χρόνο και δεν έχουν γίνει σχετικές έρευνες. Και ο νέος ε, αρχισυντάκτης έχει λάβει απειλές για τη ζωή του πριν από κάποιες εβδομάδες. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι, μιλούν από μόνα τους. Αν λοιπόν η κατάσταση μπορεί η κατάσταση να μην είναι τόσο άσχημη όσο ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή για, τους, ε, για την κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μεταβούν στις περιοχές που ελέγχονται από τους τύπους του Ταμίλ. Γιατί δεν μπορούν να μεταβούν στις περιοχές όπου πολεμήθηκε ο πόλεμος. Γιατί περιμένουν οι ξένοι ερευνητές ακόμα θεωρήσεις για να έρθουν να παρακολουθήσουν την ε, κατάσταση των εκλογών. Γιατί συνεχίζεται η προπαγάνδα υπέρ του υφιστάμενου Προέδρου. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στα κρατικά μέσα. Γιατί υποχρεώνεται κόσμος να φύγει από τη χώρα μ, λόγω απειλών. Αυτές οι απαντήσεις, αυτά τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά και επηρεάζουν Μπορεί να έχουν απελευθερωθεί, απελευθερωθεί χιλιάδες άτομα από τα στρατόπεδα εκτοπιστέντων, αλλά αυτό ήταν φυσιολογικό. Γιατί να μπουν δηλαδή οι όμοιροι σε στρατόπεδα κράτησης. Όλες αυτές οι εξελίξεις οφείλονται σε κάποια θεραλέα άτομα τα οποία παρά τις απειλές βγήκαν και είπαν τη γνώμη τους. Νομίζω ότι η έρευνα αυτή είναι πολύ σημαντική και χαιρόμαστε ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει στα σοβαρά την υπόθεση αυτή, θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις σχετικές συνθήκες. Φυσικά, όπως είπε ο πρέσβης, κάποιες χώρες τα πήγαιναν χειρότερα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως, είναι καθήκον της κυβέρνησης, είναι καθήκον της ε, σημερινής κυβέρνησης να εφαρμόσει τις συνθήκες, να σεβαστεί όλες αυτές τις βασικές θεμελιώδους ελευθερίες. Και πραγματικά οι ενδείξεις είναι ανησυχητικές. Γιατί ο πρόεδρος μετά το τέλος του πολέμου πήγε στην Βερμανία. Μα η πρώτη επίσημη επίσκεψή του διεθνής ήταν να πάει στη Βερμανία και να επισκεφτεί τον ε, στρατηγό να τον ευχαριστήσει για τη βοήθειά του. Ναι. Με το σωστό τρόπο έγινε ο πόλεμος. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεχιστεί η έρευνα αυτή και αν η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις συνθήκες θα είναι υπεύθυνη για την αναστολή του GSP Plus για τη χώρα. Ευχαριστώ. The the discussion will follow with participants. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτή τη δημόσια κρόση. About the, the, the, ε, ε, Mrs. Muscardini. Α, ναι. Η αντιπρόεδρος Μουσκαρδίνη μα ζήτησε να εκφράσουμε και τη μία θέση ως επιτροπή. Δεν έχουμε γραπτεί βέβαια, αλλά ξέρω ότι τάσετε κατά της απόσυρσης της, της ε, διαγραφής της Ρελάνκα από τον κατάλογο των γενικευμένων προτιμήσεων, διότι Εκείνη θεωρεί ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα από την τελευταία αναφορά της Κομισιόν. Λοιπόν, θα αρχίσω από τους σοσιαλιστάς και δημοκρατές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ, πολύ πολύ σύντομα. 17 λεπτά μόνο ακόμα και θα πρέπει να δοθεί ο λόγος και στην Επιτροπή και στους υπόλοιπους. Ε, από τους εξέχοντες πραγματικά ομιλητές μας. Γι' αυτό παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο ομιλία σας. Ναι, σίγουρα τέσσερις παρατηρήσεις. Ε, πρώτη, όπως υπενθυμήθηκε ακριβώς, ε, όλες οι διεθνείς εκθέσεις από διεθνή όργανα όπως κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, τι δείχνουν ότι έστω τα πολύ άσχημα κατά τη διάρκεια του πολέμου ε, και η παραβίαση των δικαιωμάτων ε, ε, διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα των πολιτών κατά τις βιοπραγίες και βασανιστήριο όλα αυτά παραβιάζονται. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και δεύτερο, η μάχη κατά των ανταρτών είναι ένα πράγμα, αλλά τώρα η καταπίεση όλων των υπολείπων, των πολιτών, των μεσόγειων κλπ. Δεν εντελώ διαφορετικό πράγμα είναι και μόνο και μόνο επειδή δίνουμε τη μάχη μας κατά τρομοσκρατίας δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε ή να πούμε ότι ναι όλα εντάξει σε όλα αυτές τις ενέργειες ε, ε, και για τους Ταμούλ και για τους δημοσιογράφους, μάρτυρες κλπ. που θέλουν να εκφράσουν την αλήθεια και ανησυχούν για όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές τις ενέργειες, τις πράξεις, ιδιαίτερα σε αυτά τα στρατόπεδα κράτησης όπου υπάρχει ιδιαίτερη απαγόρευση πρόσβασης και επίσης έχει άμεση ευθύνη το καθεστώς ο υπουργό Άμυνας που προσωπικά απειλεί, συνεχίζει να απειλεί τους δημοσιογράφους και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο αδερφός του νομίζω ότι είναι από την άλλη μεριά και εκεί σε όλα αυτά δεν μπορεί να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για ορισμένα έτσι, ατυχήματα και ορισμένες παραστατικές νάδες ε, γιατί βλέπουμε ότι καλύπτονται σίγουρα από τον ίδιο στρατό και τις επίσημες αρχές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να διατηρήσει μια πολιτική στήριξη αρχών του Σρι Λάγκα. Βέβαια μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, σίγουρα ένα διάλογο, αλλά αυτό το Ναι. Λοιπόν, το σύστημα χρειάζεται υποχρεώσεις που να γίνονται σεβαστές ε, και με ξέπληξε που άκουσα τον κύριο Γκρέι να λέει ότι η Σλάνκα ήταν της αηφόρου ανάπτυξη ένας παράδεισος. Ε, ένας μεγάλος Ευρωπαίος είπε κάτι που ήταν και συμπατριώτη σας ότι το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, ναι, κατά τον Ταμούλ να έχουμε πολιτική κάποιες λύσεις που να ε, διερευνώνται και αυτό και να αναλάβει την υποχρέωση της Λάγκα ε, να μην ε, τρομοκρατεί, να μην βασανίζει. Το ελάχιστο είναι αυτό που απαιτούμε για να μπορέσουμε να προβλέψουμε ενδεχόμενα μια καθεστώς στήριξης όπως αυτό το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Ευχαριστώ πολύ, έχουν ζητήσει το λόγο και θα πρέπει να ξεκινήσουμε και το ρολόι μας, το χρονόμετρό μας. Γι' αυτό στο εξή σας παρακαλώ Δύο λεπτά ο καθένας, μου φαίνεται λογικό. Διάν Ζάραντιλ, από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον πρέσβη και τους υπόλοιπους που μας έδωσαν τις λεπτομέρειες της κατάστασης στην Σρι Τα πράγματα είναι δύσκολα, δύσκολα ναι, αλλά Ακόμη και ο κύριος Μούσο που ήταν μεγάλος επικριτής στο λόγο του είπε ότι σε σύγκριση με αυτά που συνέβαιναν πριν από ένα χρόνο η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Αφού υπάρχει λοιπόν βελτίωση και αυτό είναι προφανές νομίζω όσο αργά και να γίνεται η βελτίωση δεν θα έπρεπε να παίρνουμε εμείς μέτρα που να χειροτερεύουν τα πράγματα και να αυξάνουν τι σημείες για τον πληθυσμό. Βέβαια έχουμε και εμείς το δικαίωμα υπό ορισμένες συνθήκες να χρησιμοποιούμε εμπορικά όπλα όπως για την επίλυση πολιτικών προβλημάτων αλλά δεν λέω ότι αυτό θα γίνει και τώρα αλλά πρέπει να ξαναδούμε να το ξανασκεφτούμε και να λάβουμε υπόψη μας και τις επιπτώσεις που θα είχαν τέτοιου είδους εμπορικά μέτρα ως προς την απασχόληση ας πούμε στην Σρι Λάγκα. και να επιδείξουμε κάποια περισσότερη υπομονή. Σας ευχαριστώ επίσης που αναφέρατε την επιστολή της Αντιπροέδρου Μουσκαρδίνη που μας διανεμήθηκε. Εγώ συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματά της και τις επικρίσεις της για την ε, διαγραφή της Σρι Λάγκας από τον κατάλογο. Νομίζω ότι με αυτό το μέτρο θα χειροτερέψουμε τα πράγματα αντί να τα βελτιώσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο Παύλος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη βούληση στην περίπτωση που δεν ισχύει πια αυτό το σύστημα να έχουμε όμως μια σταθερή συνεργασία μεταξύ ΛΑΚΑ και της Επιτροπής για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε όσο γίνεται νωρίτερα αυτό το σύστημα. Και εδώ αυτά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δόθηκε μάχη κατά της τρομοκρατίας. Έχουμε εμπιστοσύνη στη μάχη αυτή και προτείνουμε ένα έλεγχο συνεχή από πλευρά της Επιτροπής ωστόσο γίνεται νωρίτερα να επανέλθουμε στην ομαλή κατάσταση. Και ε, από τη στιγμή που θα παρατηρηθεί μια βελτίωση να προταθεί στο Συμβούλιο μια νέα πρόταση. Το Κοινοβούλιο επίσης θα ελέγχει την όλη κατάσταση, θα κάνουμε μια ανάλυση αυτής της καταστάσεως. Από τη στιγμή που σίγουρα θα βρεθεί η κατάσταση θα προτείνουμε στην Επιτροπή κάτι το καινούριο σαν πρόταση. Αυτά και πρόεδρε σας ευχαριστώ. Χωρίς προ... μικρόφωνο πρόεδρος. Σκιώδης Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και να πω ότι εξ ονόμας των Πρασίνων συμφωνώ αυτά που είπε ο Ντεζίρ για το πώς έχει η κατάσταση και τα συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να βγάλουμε. Να προσθέσω ότι για την ομάδα μου Πρώτη, εμείς υποστηρίζουμε αυτό το σύστημα γερικών προτιμήσεων ώστε οι χώρες του Νότου να αναπτυχθούν χάρη στο εμπορικές συναλλαγές. Θεωρούμε όμως ότι τα κοινωνικά τμήματα και περιβαλλοντικά σίγουρα συνδέονται με ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Για μας τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι τα δικαιώματα μέσω δημοκρατικής μάχης αγώνα και όχι των επιχειρήσεων που θέλουν έτσι με χαρά και χάρη να τους αφιερώσουν επιχειρήσεις αυτές. Τώρα ε, για την ε, μη θέση για την μη ισχύ αυτού του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Ε, εδώ διακυβεύει το λόγο και αφισβητεί το λόγο της κυβέρνησης Λαγκά και έχουμε και το λόγο της Ευρώπης που αναλαμβάνει υποχρέωση σε αυτό διακυβεύεται η αξιοπιστία μας. Χθε προχθές είχαμε την ακρόαση ενός νέου επιτρόπου και εμεί είπαμε ότι ναι, το εμπόριο μέσω του εμπορίου εξάγονται και οι ευρωπαϊκές ιδέες δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πορεία της Επιτροπής, να την υποστηρίξουμε και να έχουμε μια, ένα προσωρινό πάγωμα μέχρι να βρεθεί η κατάσταση. Προσωρινό πάγωμα λοιπόν του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Ζων Χίγγενς από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κανένας, απολύτως κανένας δεν θέλει να δημιουργηθεί μια κατάσταση κατά την οποία θα αυξηθούν τα προβλήματα των απλών εργαζομένων και των πτωχών στην Σρι Λάγκα. Καθόλου και μάλιστα. Αλλά η κυβέρνηση θα φέρει την ευθύνη εάν ληφθεί μια απόφαση να φύγει η Σρι Λάγκα, να της αφαιρεθεί το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων. Εκείνη θα πταίει για τις παραβιάσεις που έχει κάνει και στο παρελθόν αλλά όπως ακούσαμε σήμερα και για τη συνέχιση των παραβιάσεων των πολιτικών δικαιωμάτων του λαού της και Ταμίλ και συγκάλα και δημοσιογράφους και αντιφρονούντες. Και εμείς αυτό ακούμε τι παθαίνουν, τι υφίστανται οι απλοί άνθρωποι. Και στις περιπτώσεις εμπορικών συμφωνιών με άλλες υπήρους και χώρες, αυτό μας ενδιαφέρει πάντοτε οι απλοί άνθρωποι και η μοίρα τους. Και φυσικά έρχονται εδώ εκπρόσωποι της κυβέρνησης και μας λένε παραμύθια περί ιδεωδών καταστάσεων. Αλλά αυτά είναι απλώς ψευδή. Και εμείς δεν πιστεύουμε την κυβέρνηση λόγω του παρελθόντος της. Ο λαός μπορεί να έχει επιλογή αλλά και οι δύο υποψήφοι ήταν μέχρι το λαιμό βουτυγμένοι στη σύραξη. Εναλλακτικές προτάσεις ακούγονται αλλά δεν έχω φτάσει μέχρι τις κάλπες. Και δεν αρκεί κύριε Πρόεδρε, δεν αρκεί να λένε ορισμένοι «Α, μα αφού έχει βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση, ας μας ικανοποιήσει αυτό». Εμείς θα ήμασταν ικανοποιημένοι σε μια χώρα όπου συνεχίζονται τέτοιου είδους παραβιάσεις. Δεν, δεν αρκεί αυτό. Ο εκπρόσωπος της ομάδας των φιλελεύθερων. Πρόεδρε, ευχαριστώ μπερδεμένος είμαι με τη συζήτηση αυτή. Πολλά, πάρα πολλά στοιχεία εμφανίζονται που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες συζητήσεις και χρειάζεται μια κάποια... Ε, έχουμε ως μεσαφερίες και επιφυλάξεις ε, εδώ οι εκθέσεις για τη Στριλάνκα δεν έχουν ε, την ίδια μορφή και σήμα από την Crisis Group που είναι πραγματικά σοβαρή οργάνωση δείχνει την σκληρότητα του καθεστώτος της Ρλάνκα αλλά και ορισμένα στοιχεία θετικά αναγνωρίζει σαν τάση τουλάχιστον και αυτό θα πρέπει να τα εισακούσουμε. Όταν λέει ότι είναι αρνητική η εικόνα της Λάγκα, αλλά οι προοπτικές είναι θετικές ε, στα βήματα τουλάχιστον προς μια βελτίωση της καταστάσεως, νομίζω ότι αποτελεί ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν να πάρουμε αποφάσεις για τιμωρίες. Ε, η, επι... Ε, η στάση της Επιτροπής με απόφαση τρομερά γοργή όταν τιμωρείται εμπορικά μια χώρα και όχι μόνο με αυτό το σύστημα γενικών προτιμήσεων ε, αυτό γίνεται πάντα με ιδιαίτερη επιφύλαξη, ακροάσει, διαβουλεύσει, επαφέ κλπ. Ο προηγούμενο επιτροπού Αστων η απόφαση λήφθηκε τρομερά γρήγορα. Και σήμερα εδώ δεν είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων χρησιμοποίησαν άλλοι για βρετανική ενδοσυζήτηση. Βρετανός ο Επίτροπος, βρετανικές οι παρεμβάσεις προς τη μέση κατεύθυνση μια ιδιαίτερη ε, επίσης συμμετοχή των Ταμίλ στη Μεγάλη Βρετανία που εμπόδισαν μια αντικειμενική ανάλυση καταστάσεω και τέταρτο, όταν λέμε εμεί ότι θα πρέπει να μα χαρακτηρίζει μια στάση με συνοχή όπω και απέναντι σε άλλε χώρε, είναι κάτι αληθινό. Δεν είναι απλά και μόνο μια δικαιολογία. Παρακαλώ, σεβαστείτε το χρόνο σα, λέω πρώτα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, θα ολοκληρώσω τάχιστα και σε λίγο πάω στην Λωρίδα της Γάζας και εκεί οι ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής ε, η πολιτική μας είναι πολύ πιο ανεκτική σε σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα απέναντι στη Στριλάνκα Να πω κάτι τελευταίο ολοκληρώνω. Το σύστημα κοινωνικών υποτιμήσεων είναι κατά των εργαζομένων από ό,τι γνωρίζω εγώ. Δεν είναι μια βοήθεια άμεση από όρισμε κοινωνήσει με την υποστήριξη του προπολογισμού όπω το κάνουμε στι Αφρικανικέ χώρε. Γι' αυτό παρακαλώ ιδιαίτερη επιφύλαξη. Η Επιτροπή νομίζω ότι Μιλάμε για την απόφασή της τους επόμενους έξι μήνες ακριβώς που θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε για να εφαρμοστεί η απόφαση ο νέος επίτροπος όλοι μας θα μπορέσουμε να αναλύσουμε καλύτερα και πιο ισορροπημένα την κατάσταση του θέματος. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα όλους που λέγονταν τον λόγο και τους συναδέλφου επίσης. Λοιπόν, θα πω τα εξή. Συστάθηκε μια επιτροπή έρευνα, το επιθύμησε ο Ρλεμ, ε, για τρία σημαντικά θέματα. Πρώτα απ' όλα για τι αρχέ, τι αξίε, τουλάχιστον σε παγκόσμια κλίμακα. Και η δισημενή διαπίστωση ποια είναι. Ε, υπάρχουν βήματα θετικά το γνωρίζουμε Αλλά τα πράγματα, αυτά τα βασανιστήρια δικαιώματα των πολιτών και των παιδιών, ότι γίνονται σεβαστά αυτά, είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Ακόμα ένα δεύτερο στοιχείο Σαν Ευρωπαίοι εμείς, και εντάξει, εγώ δεν είμαι υποχρεωτικά υπέρ των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, μιλάω για τους συναδέλφους εδώ. Εάν υποστοδρομήσουμε, επιστοχωρήσουμε εμείς ε, Κάθε φορά που πιστοχωρούμε επειδή υπάρχουν διάφορα συμφέροντα για τους παραγωγούς μας ή για τους καταλατές μας ε, που είναι ε, οι αρχές όμως είναι παγκόσμιου χαρακτήρα τότε να το κόψουμε ε, να μην έχουμε έτσι να μην λέμε μεγάλα λόγια, φραστικά πυροτεχνήματα κλπ γιατί κανείς να με πιστεύει πια σε παγκόσμια κλίμακα αν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κυρώσεις από τη στιγμή που δικαιολογούνται παρόμοιες κυρώσεις και ακόμα ένα τρίτο που χαρακτηρίζει την όλη σκέψη μου με... Δεν είναι καθόλου θετικό για μένα, έστω και αν δεν σημαίνουν πράγματα που λέγονται και από τον κύριο Γκρέι και ορισμένου συναδέλφου που θεωρούν ότι η ευτυχία των καταναλωτών και των μηχάνων των Ευρωπαίων θα πρέπει να πληρώνεται με αίμα ανδρών γυναικών σε ορισμένε χώρε τη Ευρώπη. Είναι εντελώ απαράδεκτο αυτό για μένα. Έτσι. Αυτό με σοκάρει λοιπόν. Ε, ζούμε σήμερα σε μια φάση που τώρα θα ληφθεί μια απόφαση και έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα και για έξι ολόκληρους μήνες ε, έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε, να αναθεωρήσουμε την απόψή μας και την απόφασή μας. Ε, είναι η ευκαιρία για τη Σλάνκα να αποδείξει ότι βελτιώνεται η κατάσταση εκεί και τότε, μόνο τότε θα μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε αυτή την απόφαση την, για να ισχύσει και πάλι το σύστημα αυτό για αυτή την περίοδο. Κύριος Κασπερή από το ΕΛΚ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η κατάσταση στη Σρι Λάγκα δεν είναι σαφώς τόσο ιδανική όπως ε, η κατάσταση την οποία φανταζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να σκεφτούμε το εξή. ακόμα και αν δεν είναι ιδανική η κατάσταση εκεί, τι μέτρα θα πάρουμε, ποιον θα πλέξουμε με τα μέτρα αυτά. Όπως είπε ο συνάδελφος, δεν θα πλέξουμε την κυβέρνηση πρωτίστως, αλλά τους πολίτες, τον κόσμο που ζει στη χώρα, που εργάζεται στη χώρα και που μπορεί να χάσει τη θέση την εργασία τους. Δεν μιλάμε για τον πρόεδρο, μιλάμε για τον κόσμο που πρέπει να βγάλει το ψωμί του. Νομίζω λοιπόν ότι γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά να μην χρησιμοποιούμε μέτρα τα οποία δεν εφαρμόζονται πουθενά άλλου. Συμφωνώ υπάρχουν πάρα πολλές χώρες τις οποίες δεν τηρούνται τα δικά μας πρότυπα, αλλά ας κοιτάξουμε τι γίνεται με την Κίνα και τις εμπορικές μας σχέσεις. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και υπάρχουν αναρρύθμιτα άλλα τέτοια παραδείγματα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τυχάνουν του σεβασμού που θα θέλαμε. Αλλά θα... δεν διακόπτουμε τις εμπορικές σχέσεις μαζί τους γι' αυτό. Να αποτρέψουμε λοιπόν αυτό που είπε ο συνάδελφος Γναλτίνη, δηλαδή τα θέματα, τα εσωτερικά πολιτικά της ε, Βρετανίας, για παράδειγμα, να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχουμε και έξι μήνες στη συνέχεια στη μεταβατική φάση. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το χρόνο αυτό για να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη θέση του και προκειμένου να επηρεάσουμε και την απόφαση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι διαμόρφωσαν και ήταν σαφές από τα σχόλια των συναδέλφων ποια είναι η γενική κατεύθυνση των σχολείων του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε την ανταλλαγή απόψεων για τη Σιρλάνκα, θα δώσω το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρία λεπτά. Μετά από τα νέα στοιχεία που μας μετέφερε ο πρέσβης της Σριλάνκα. πιστεύετε ότι μπορούμε να αναθεωρήσουμε τη θέση μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω κι εγώ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή συζήτηση. Καταρχήν θα ήθελα να επαναλάβω ε, κάτι που είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρία όταν παρουσιάσαμε στις 10 Νοεμβρίου το θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα πορίσματα της διερευνητικής έκθεσης. Αυτή ήταν και η βάση για τα βήματα που έλαβε ε, και τις προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα αυτή ήταν ε, το πέρας μιας χρονοβόρας και διεξοδικής διαδικασίας που έλαβε υπόψη όλα τα υλικά και τα στοιχεία που λάβαμε και από τη Σρι Λάνκα και από άλλες διάβλους Πάντως ήταν, επαναλαμβάνω, ε, κατακλείδα μιας ε, μακροχρόνιας ε, ερευνητικής προσπάθειας. Σε καμία περίπτωση δεν θελήσαμε να επισπεύσουμε τα πράγματα. Με βάση λοιπόν αυτές, αυτά τα πορίσματα υποβάλαμε στο Συμβούλιο μια πρόταση για προσωρινή απόσυρση. Αν εγκριθεί η πρόταση αυτό το Συμβούλιο θα τεθεί σε ισχύ μετά από 6 μήνες. Επίτηδες έχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, αυτή την προθεσμία προκειμένου να προλάβουν οι χώρες να αναλάβουν ε, δράσεις να διορθώσουν το πρόβλημα και να διασκεδάσουν τις ανησυχίες που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία. Δεν θέλουμε να δείξουμε ότι ε, σπέβδουμε να άρουμε τα πλεονεκτήματα του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Θα ήθελα να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι το μέτρο αυτό δεν είναι επουδενή μέτρο προστατευτισμού. Αν συμφωνήσει το Συμβούλιο με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ισχύσει η απόσυρση, η Σρι Λάγκα θα επανέλθει στο κανονικό σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και θα υπάγεται στου ίδιου κανόνε και στην ίδια πρόσβαση με του υπόλοιπου εταίρου στην περιοχή. Αυτή, αυτή τη στιγμή έχει καλύτερη πρόσβαση λόγω του ΣΥΝ, των γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, γιατί μέχρι στιγμή ε, εκπλήρωναν τι προποθέσει αυτού του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, που είναι ένα είδο διαπραγμάτευση ε, με προνομιακού εταίρου Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όταν δεν τηρούνται οι αμοιβέ υποχρεώσεις λαμβάνονται και κάποια μέτρα. Δεν είναι αμυροσυνεπιών με μια τέτοια θέτηση υποχρεώσεων. Έχουμε συχνό διάλογο με εκπροσώπους στη Σρι Λάγκα και μακάρι να στοιχειοθετηθεί μια νέα πρόταση για την επαναφορά στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε τη διαβεβαίωση για αυτά μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση της Σρι ώστε να βελτιωθεί το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο της χώρας αυτής και να διορθωθούν τα προβλήματα και εγκατασταλείς που διαπιστώθηκαν στην διερευνητική έκθεση. Πάντως σας βεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στο θέμα και θα συνεχίσει το διάλογο με την κυβέρνηση της Σρι και θα χρησιμοποιήσει και άλλες διάβλους. Και αν καταφέρουμε... Ολοκληρώστε παρακαλώ γιατί ξεπεράσετε το χρόνο σας. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε αλλαγή της κατάστασης θα επανυποβάλουμε πρόταση για επαναφορά της Ριλάνκα στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Καλώς, ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Και αυτή τη φορά θα αρχίσω με τον κύριο Ζένον τον Διεθνή Συντονιστή της Αλληλεγγύης Ταμίλ. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επαναλάβω ορισμένα από τα στοιχεία που σας έδωσα προηγουμένως. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ε, κυβέρνησης της Σρι και κάποιων ε, μελών της Επιτροπής είναι ότι η άρση αυτή θα επηρεάσει τους εργαζόμενους που εποφελούνται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝΑ. Αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται προς όφελος των εργατών. Ιδιαίτερα των εργαζομένων στην φαντουργία ή στη βιομηχανία ε, Σε παραλαμβάνω η βιομηχανία αυτή έχει καταστραφεί από το στρατό και δεν έχει αποκατασταθεί. Τα χρήματα ε, ενθυλακώνονται από κυβερνητικούς παράγοντες και εξυπηρετούν ουσιαστικά την διαφθορά. Και γίνονται κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση της Σριλάνκα. Ε, τα στρατόπεδα κράτησης ε, είναι χειρότερα και από τα στρατόπεδα της Παλαιστίνης. Είναι τελείως απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν και θα ήταν κολοσιαίο λάθος για οποιοδήποτε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και που διεκδικεί βελτίωση του επίπεδου ζωής των φτωχών αυτών ανθρώπων να εγκρίνει ε, μια τέτοια πρόταση για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Μία τέτοια λύση θα ήταν ουσιαστικά προδοσία των, ε, ε, θεμελίων του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή της κατάστασης, η ε, ομάδα για τη διεθνή κρίση έχει συντάξει έκθεση για το πώς αλλάζει η κατάσταση, αλλά 150.000 άνθρωποι μέσα σε δύο εβδομάδες το Δεκέμβριο απελευθερώθηκαν μετά την διακήρυξη της ημερομηνία των εκλογών και μετά την τη δήλωση του Φονσέκα ότι θα κατέβει στις προεδρικές εκλογές. Είπε ότι Έκανε λοιπόν αυτές τις δηλώσεις και υποσχέθηκε απελευθέρωση 150.000 κρατουμένων. Βέβαια υπάρχουν ακόμη κέντρα κράτησης, που δεν τα λένε κέντρα κράτησης, αλλά κέντρα διαμετακόμισης. Παρ' όλα αυτά όλα είναι προεκλογικές υποσχέσεις. Στην πράξη τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ούτε πολιτική λύση διαφαίνεται, ούτε καμία προσπάθεια αποκατάστασης. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο ότι θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης στις πληγήσεις περιοχές. Και το θέμα της ε, καθάρισης από τις ενάρκε. Εκεί ζούσαν άνθρωποι. Ε, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε χωριά που είναι ναρκοπαίδια. Ολοκληρώστε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυβέρνηση είπε ότι θα κλείσει όλα τα ειδικά κέντρα και στρατόπεδα κράτησης. Αυτό πρέπει να το κάνει όμως, όχι μόνο λόγια. Έχουμε και δεκάχρονα παιδιά που κρατούνται σε τέτοια κέντρα. Και ο πρέσβης της Σρι έχει άλλο ένα τρίλεπτο για να απαντήσει. Θεωρείτε ότι είναι παρκή τα τεκμήρια που προσκομίσατε προκειμένου να αποδείξετε την αλλαγή της κατάστασης. Όπως είπε και στην αρχή και τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό προς την Επιτροπή σας. Εγώ δεν είπα ότι η Σρι δεν έχει προβλήματα. Ήταν σαφές αυτό. Αλλά σας επισήμανα το πλαίσιο στο οποίο έλαβα χώρα όλα αυτά. Το πλαίσιο αυτό έχει αλλάξει, έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση, οπότε μπορούμε να επανέλθουμε σε πιο ομαλές συνθήκες. Ο εκπρόσωπος των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα επισήμανε και αυτός κάποιες βελτιώσεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Και διαπιστώνω ότι το αναγνωρίζουν και κάποιοι ευρωβουλευτές. Και οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να αναγνώρισε αυτή τη βελτίωση. Ποιο είναι αυτό το μαγικό κατόφλι για την ε, έμπρακτη ή αποτελεσματική εφαρμογή. Αυτό θα πρέπει να προσδιορίσουμε. Είναι σημαντικό, εκτός από την αλλαγή, ό,τι κάνετε προς τη Σρι να είναι ισότιμο με αυτά που εφαρμόζεται για τους υπόλοιπους εταίρους του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Αλλιώς παραβιάζεται τις προδιαγραφές και απαιτήσει της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Σας απευθύνω λοιπόν έκκληση να λάβετε σοβαρά υπόψη αυτό το γεγονός. Δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση και είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σύγχυση ως προς την α, λήψη της απόφασης. Αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για πολύ πιο ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης. Ξανασκεφτείτε το λοιπόν, σας θερμό παρακαλώ, δώστε ακόμη, λίγο ακόμη χρόνο στη Σρι για να ανασκουμποθεί και να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό θα ικανοποιήσει και τους κυρίους Αρίφ και Ντεζίρ και τον κύριο Ζαντό. Αλλά δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε κάποιου που αδιαφορούν για την επίλυση του προβλήματος. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτού που είναι λογικοί και χέφρονες και θέλουν πραγματικά ένα αποτέλεσμα. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω και την απογοήτευσή μου από τον εκπρόσωπο του Ταμίλ, ε, αλληλεγγύη του Ταμίλ. Όλα αυτά που είπε ήταν κλισέ στερεοτυπίες και γενικότητες. Εγώ σα έδωσα συγκεκριμένες πληροφορίες, σας έδωσα στατιστικές που έδειξαν την ε, εμφανή βελτίωση φέτος. Δώστε μου κι εσείς στοιχεία που να διαψεύδουν τα στατιστικά που σας παρουσίασα. Δεν χρειάζεται καν να, να απαντήσω. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Η διασπορά της ε, Σριλάνκα έχει διεκδικήσεις που μερικές φορές είναι άσχετες από τις απαιτήσει του λαού της Σριλάνκα. Δεν θα πρέπει οι άνθρωποι που μένουν εκτός της Σρι να καθορίζουν την τύχη της. Αφήστε τους ανθρώπους Σρι να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψε. Και χαίρομαι που είχαμε προγραμματίσει αυτή την ακρόαση. Δείχνει το πόσο ανοιχτό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πόσο ανοιχτό μυαλό και φέρνει διστάμενες απόψεις στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και τα συζητούμε όλα και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Move to point 10 of our... Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διατάξη, στο 10, συμφωνία σχετικά με το εμπόριο μπανάνας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προμηθευτών μπανάνας και έχουμε μαζί τον κύριο Σάλιβεν από τη Γενική Διεύθυνση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και καλώς ορίσατε. Οι δερμηνείς θα μείνουν μαζί μας για μισή ώρα ακόμα τουλάχιστον. Τουλάχιστον για να ανακληρώσουμε την συνεδρίαση στη μία, αν χρειαστεί, τονίζω. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Δεκέμβριο, τον Περσινό, λίγο μετά τη συνάντηση κατά την οποία συζητήσαμε το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής κατέληξαν σε μια συμφωνία για τους δασμούς, κλείνοντα μια, κλείνοντας μία από τις πιο μακροχρόνιες διαμάχες για τέτοιο εμπορικό θέμα. Ο Πασκάλ Νταμή είπε ότι επρόκειτο για ένα από τα πιο περίπλοκα πολιτικά ευαίσθητα θέματα τα οποία έχουν ε, τύχει διαπραγμάτευση στον ΠΟΕ. Με τη συμφωνία αυτή Εισάγονται πολλοί τόνοι φρούτων κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς. Πολλές χώρες λοιπόν της Λατινικής Αμερικής στις οποίες συγκαταλέγονται και κάποιοι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μπανάνας θεωρούν ότι γίνεται διακριτική μεταχείριση υπέρ των προϊόντων από τις χώρες ΑΚΕ και ότι παραβιάζονται οι κανόνες σχετικά με τους ε, περιορισμούς ω προς τον όγκο. Ο ΠΟ υποστήριξε τις ε, κατηγορίες αυτής και αναθεώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα περιορίσει τους δασμούς της σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές μπανάνας από χώρες ε, Λατινικής Αμερικής από 115 ευρώ ανατόνο το 2017 με, μάλλον στα 115 ευρώ ανατόνο το 2017 και η, μπανάνα από τις χώρες ΑΚΕ θα συνεχίσει να εισάγεται χωρίς δασμούς με τα ειδικά πλεονεκτήματα. Οι βασικές χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνα θα λάβουν ως 200 εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια προκειμένου να προσαρμοστούν στην μείωση των πλέον εκτιμάτων τους. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Οσάλιβαν, Γενικό Διευθυντή της Διευθυνσής Εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας παρουσιάσει την συμφωνία και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο και για το γύρο της Ντόχα, αλλά και για τις χώρες, τις εμπλεκόμενες. Σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να ενημερώσω την Επιτροπή ότι μετά την τελευταία μας συνάντηση πριν από τα Χριστούγεννα σας είχα πει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει συμφωνία όπως και έγινε και αυτό ήταν απάντηση σε τρία σε τρεις εντολές. Καταρχάς μία νομική εντολή γιατί μας είχαν καταδικάσει διάφορα πάνελ του ΠΟΕ και δεν ε, συμβαδίζουμε ακόμα αν θέλετε, δεν συμμορφωνόμαστε με τις αποφάσεις ε, των εμπορικών διατάξεων ε, του ΠΟΕ. Κατά δεύτερον είχαμε μία διαπραγματευτική εντολή γιατί αν δεν είχαμε διαπραγματευτεί ένα ειδικό καθεστώ για την μπανάνα δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το γύρο τη Δόχα γιατί δεν θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε την μεταχείριση της μπανάνας ως τροπικό προϊόν. Καταλαβαίνω ότι είναι κάπως αντιφατικό το επιχείρημα αυτό γιατί η μπανάνα είναι το πλέον τροπικό από όλα τα προϊόντα κατά πάσα πιθανότητα αλλά από οικονομική άποψη μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε να βρεθεί μια ξεχωριστή ένας ξεχωριστός τρόπος αντιμετώπισης της μπανάνας και ύστερα η ανάγκη να συναυτεί μια συμφωνία γενικά για τα τροπικά προϊόντα, όπου και πάλι είχαμε μια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί υπήρχε φυσικά συμφέρον από πλευράς Ευρωπαίων παραγωγών να μην ε, χαρακτηριστούν κάποια συγκεκριμένα προϊόντα ως τροπικά προϊόντα και φυσικά υπήρχε και το συμφέρον για τις χώρες ΑΚΕ σε ό,τι αφορά την διάβρωση των προνομίων τους γιατί δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία για τις μπανάνες και τα τροπικά προϊόντα χωρίς να συμφωνήσουμε και πώς θα αποζημιωθούν οι ναι, χώρες. ακέ ναι. από... σε σχέση με την διάβρωση των προνομίων τους. Αυτά λοιπόν ήταν τα στοιχεία που μας απασχολούσαν. Και τέλος, όπως είπα, είχαμε και μια πολιτική αλλά και ηθική, αν θέλετε, επιταγή να προσπαθήσουμε μια και καλή, να αφαιρέσουμε αυτό το δηλητηριώδες, αν θέλετε, θέμα από τις διαπραγματεύσεις μας, το οποίο μας κοστίζει πολλά στις διαπραγματεύσεις μας και διαβρώνει πολύ τη φήμη μας και στη Γενέβη και ανακύπτει σε πάρα πολλά βήματα. Νομίζω ότι όλοι αναγνώρισαν ότι έπρεπε να βρεθεί μια οριστική λύση. Το πετύχαμε λοιπόν τώρα αυτό. Ε, πρόεδρε, τώρα ό,τι μου πείτε σε σχέση με το χρόνο, δεν προτείνω. Εκτός και αν θέλετε να υπησέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες, δεν προτείνω να το κάνω αυτό. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε πλέον στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα πρότεινα σε άλλες συνθήκες να κάνουμε μια τεχνική συνάντηση για να παρουσιάσω τις ε, λεπτομέρειες, αλλά δεν ε, έχουμε τον ίδιο μηχανισμό πλέον. Θα είναι χαρά μου όμως να σας κάνω μια τεχνική ενημέρωση για τους βοηθούς, για τα μέλη του Κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται, αλλά ίσως όχι σήμερα γιατί είναι πολύ χρονοβόρα αυτή η διαδικασία, αλλά νομίζω είναι σημαντικές οι λεπτομέρειες. Αν θέλετε λοιπόν, ευχαρίστω να οργανώσουμε μια τέτοια ενημερωτική συνεδρίαση για όσους ε, ενδιαφέρονται. Για να καταλάβει και το Κοινοβούλιο τον τεχνικό αντίκτυπο, την νομική δομή Τη συμφωνία. Γενικά, αφενό τι έχουμε. Μία συμφωνία για την μπανάνα. Για την επίλυση της, ε, των διαφορών που ορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης της μπανάνας στα πλαίσια του γύρου της Δόχα ή και εκτός του γύρου της Ντόχα για την ε, επιτεύξη των περικοπών. Αυτό σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές από τη Λατινική Αμερική. Εκ παραλλήλου έχουμε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία δεν είναι ένα τέλος στη διαμάχη που υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ορίζει και τους σχετικούς όρους. Επίσης ένα πακέτο για τα τροπικά προϊόντα και για την διάβρωση των προτιμήσεων. Στην περίπτωση της διάβρωσης των προτιμήσεων είναι δημόσιο ο κατάλογος για τα την διάβρωση των προνομίων δεν είναι δημόσιο ο κατάλογος. Τα κράτη-μέλη όμως έχουν ενημερωθεί πλήρως σε ό,τι αφορά τον κατάλογο αυτών των τροπικών προϊόντων και νομίζω ότι έτσι προστατεύονται τα συμφέροντά μας από αυτή την άποψη. Και τέλος έχουμε και μία ξεχωριστή συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό προσαρμογής της μπανάνας και σας υπόσχομαι ότι δεν θα αναφερθώ ποτέ στο μηχανισμό αυτό με το αρκτικό λέξό του. για να προσαρμοστούμε, να προσαρμοστούν οι χώρες αυτές στις νέες εμπορικές καταστάσεις, συνθήκες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό το πίσω και να αφορά πιο έντονα το Κοινοβούλιο εδώ και τώρα σήμερα, καταρτίζουμε τα νομικά κείμενα στην παρούσα φάση, τα οποία και θα παρουσιαστούν στο Σώμα των Επιτρόπων ε, το συντομότερο δυνατόν. Φυσικά δεν γίνεται αυτό να τα παρουσιάσουμε στην Υπηρεσιακή, Κυβέρ... στην Υπηρεσιακή Επιτροπή. Θα πρέπει να περιμένουμε το διορισμό της Επιτροπής. Ξέρω ότι διεξάγονται Συζητήσει οι οποίες γίνονται σε πολιτικό επίπεδο. Μετά θα ζητήσουμε από το πολιτικό, από το Συμβούλιο των Υπουργών να εγκρίνει την απόφαση και να την υπογράψει. Και φυσικά θα τηρήσουμε το Κοινοβούλιο απόλυτα ενήμερο. Από τη στιγμή που θα έχει υπογραφεί η συνθήκη θα έρθει στο Κοινοβούλιο για έγκριση, γιατί φυσικά πρόκειται για διεθνή συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία έχουμε δύο τμήματα όπου θα ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις. καταρχά σε ό,τι αφορά τον, ε, το τροποποιημένο τέλος. Θα αρχίσουν δηλαδή ήδη περικοπές και ύστερα η ρήτρα δέσμευσης και για τα δύο μέρη ότι δεν πρόκειται να, να κινηθούν να κινηθούν νομικές διατάξεις όσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συμφωνία. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην παρούσα φάση ε, θα εφαρμοστούν προσωρινά αυτές οι δύο πτυχές και αν τυχόν το Κοινοβούλιο καταψηφίσει τη συμφωνία θα πάυσουν να ισχύουν αυτές οι προσωρινές διατάξεις και θα επιστρέψουμε στους αρχικούς δασμούς. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα και θα πρέπει να συζητηθούν και με την ε, Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε σήμερα. Μία μικρή παρένθεση, επιτρέψτε μου. Αυτή η συμφωνία είναι, αν θέλετε, χαρακτηριστική ως προς τη φύση της ε, σε σχέση και με κάποιες άλλες ε, συμφωνίες που θα ακολουθήσουν, που δεν είναι πολύ ευρείες, αλλά είναι διεθνείς συνθήκες στα πλαίσια της συνθήκης. Άρα, χρειάζεται το ενδιαφέρον σας, αλλά δεν είναι μεγάλες ε, διεθνείς συνθήκες. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί το διαδικαστικό σκέλος. Γιατί δεν θέλουμε να βαρύνουμε και να καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Δεν έχω υπόψη μου κάποια απόλυτη λύση. Έχουν ξεκινήσει συζητήσει με την γραμματεία και υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να περάσουν από την έγκρισή σα, αλλά υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί και περιορισμοί ω προ την μεθοδολογία. Άρα θα πρέπει να δούμε πώ θα διασφαλίσουμε ότι ναι, μεν είσαστε σε θέση να ασκήσετε τις, τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει που προβλέπει η συνθήκη, αλλά παράλληλα θα είμαστε και σε θέση να προχωρήσουμε τι διαπραγματεύσει στη Γενέβη για τι συμφωνίε αυτέ. Το πακέτο υποστήριξη των ΑΚΕ θα είναι ξεχωριστό νομικό εργαλείο που θα τροποποιεί ένα από τα υφιστάμενα μέσα για παροχή βοήθειας και αυτό θα περάσει από συναπόφαση φυσικά. Θα ολοκληρώσω λοιπόν στο σημείο αυτό. Θα έχετε και ερωτήσεις φαντάζομαι, αλλά αν θέλετε να διοργανώσουμε κάποια καλύτερη στιγμή μια τεχνική συνάντηση για να εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες προκειμένου να έχει την αίσθηση και η Επιτροπή σας ότι είναι απόλυτα ενημερωμένη για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Και φυσικά να επανέλθουμε σε μετέπειτα επιταφάσεις, σε συζητήσεις. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη πολιτική αξιολόγηση του θέματος, λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε σίγουρα στο μέλλον στο θέμα αυτό. γιατί μπορεί να χρειαστεί και να το εγκρίνουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ λογική και σωστή η πρόταση που έκανε ο Γενικός Διευθυντής Ντέβιλ Σάλιβαν για την διοργάνωση μιας συνάντησης τεχνικών στοιχείων όχι μόνο με τους βουλευτές αλλά και τους πολιτικούς φορείς και ίσως και τους βοηθούς των ε, βουλευτών. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμος ο τρόπος αυτός για να βοηθηθούμε, να ενημερωθούμε ναι, ναι, ναι. για τη συμφωνία αυτή. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Κάντερ Αρή. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε πίεση χρόνου και να είστε σύντομοι. Δύο λεπτά. Ο Κάντερ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επανέλθω στο θέμα της ίδιας συμφωνίας, έστω και αν διαπιστώνουμε υποχρεωτικά, όπως τα έκανε ο Φεροβάλλον και ο κ. Δεγκούχτ, ε, στην επιστολή του τέλος Δεκεμβρίου, στο συνοηστή το χρόνο και για την Μπανάνα, ε, υπουργό του Καμερούν ε, να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, όχι μέρος του σε όλη συζήτηση, αλλά με απασχολεί 100 εκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, 2010-2013 για αυτή την περίοδο λοιπόν. 200-200 εκατομμύρια, στην αρχή ήταν 250 εκατομμύρια, αρκετά σημαντικά για αρκετές χώρες, αλλά πίσω από αυτό και ακούστηκε ήδη δεν είναι να βοηθούν όλες οι χώρες. Ποιες είναι οι χώρες που βοηθούνται από τις χώρες ΑΚΕ για αυτά τα 200 εκατομμύρια. Όλες οι χώρες που παράγουν ή μόνο η μεγαλό παραγωγή μπανάνας δεύτερη τώρα παρατήρηση και μετά το 2013 θα ισχύσει αυτή η ενίσχυση. Τρίτο ερωτηματικό, η βοήθεια αυτή ε, μέσω του προπολογισμού θα πάει άμεσα στους παραγωγούς είτε θα περάσει από κυκλώματα κυβερνητικά και χωρίς υποχρεωτικά να υπάρχει και η απαραίτητη διαφάνεια ε, και η βοήθεια ακριβώ για τους παραγωγούς που εκείνοι τη χρειάζονται. Και ακόμα κάτι στα κείμενα λέτε ότι σίγουρα χρειάζεται μια διαφοροποίηση και ε, κάτι το σύγχρονο, αλλά πώς, με ποια μέσα θα γίνουν αυτός ο εξυγχρονισμός και, το, και πώς αποτελεσματικά θα είναι επίσης συμπληρωματικά καλύψει μέσω του ΦΕΔ, αλλά εδώ έχουμε μόνο 4% του συνολικού ποσού ανάπτυξη. Τίποτα για τα ολοκληρωμένα περιφερειακά προγράμματα, πολύ λίγα. Εντάξει, με εκπλήσει λοιπόν κάπω το πράγμα και επειδή ήμουν εισηγητή για την Κεντρική Αφρική, για το Καμερό συγκεκριμένα, στην περιφερειακή στρατηγική, στο έγγραφο αυτό για την Κεντρική Αφρική δεν υπήρχε τίποτα που να συμπεριλαμβάνεται και ειδικότερα για το Καμερούν που είναι και ο μεγαλύτερο παραγωγό μπανάνα. Τελευταίε λέξει τώρα προβλέπεται μια κάποια ενίσχυση και με συγχωρείτε, σαν Ευρωπαίοι, εμεί νομίζω ότι μας αφορά το θέμα για τις υπερπεριφερειακές ε, ε, περιοχές ε, βάσει ποια στήριξης, με ποιο τρόπο. Ευχαριστούμε τον Γκαντέρ Σάλβα από το ΕΛΚ. Πάουλ Σάλβα. Ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εδώ τελικά ε, είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και πέρασαν περίπου 20 χρόνια για να πετύχουμε αυτή τη συμφωνία και νομίζω ότι αποτελεί ε, κάτι το πολύ σημαντικό εδώ και ε, βέβαια θα πρέπει στις συνεργασίες για την Τόχα είναι και με ιδιαίτερη έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα. Θα ήθελα ακόμα κάτι να πω, να τονίσω ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μπανάνας οι περισσότεροι βρίσκονται σε, περ, σε όπω περιοχές όπως τη Μαδέρα ή στα Κανάρια νησιά. Δεν θέλουν έτσι αυτόν τον τρόπο για το μέλλον και όπως το είπαμε και το είπαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά και ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Παύλο. Και τώρα ποιος? Γιάννη Ξαντού. Γιάννη Ξαντού. Ε, ε, ναι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το θέμα αυτών των προγραμμάτων στήριξης σε αυτή τη μεταβατική περίοδο είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και μιλάμε με οικονομικούς όρους και νομίζω ότι δύσκολο, περίπλοκο είναι να ξέρουμε τελωνιακά έσοδα που έχουν να κάνουν με την μπανάνα. Τι γίνεται με αυτά διαθέτουμε στατιστικές για να γνωρίζουμε ακριβώ ε, γιατί αυτά τα χρήματα των καταναλωτών ε, σε ποιους πάνε και τι, με τι ποσά έχουμε να κάνουμε γύρω από τελωνιακά τέλη κλπ. Ε, για την εισαγωγή μπανάνας, τι γίνεται και γραπτός σε αιτήσια βάση μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία αυτά. E. Ο Τζο Higgins από την ΚΟΕ. E. Ευχαριστώ. Τρεις σύντομες ερωτήσεις προς τον κύριο Σάλιβαν. Στο προηγούμενο καθεστώς, κύριε ο Σάλιβαν, υπήρξαν αρκετές εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και των παραδοσιακών χωρών παραγωγής και αντιδικής και μεταξύ των εταιριών. Ποια ήταν η δράση, η στάση των χωρών ΑΚΕ σε σχέση με τη νέα συμφωνία. Ποια είναι η θέση τους. Η Ονδούρας είναι σημαντικός εξαγωγές μπανάνας. Βέβαια, έχουμε μια δύσκολη πολιτική κατάσταση και την εκλεγμένη κυβέρνηση να έχει ανατραπεί από μια δικτατορία. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία, εκπρόσωπος των πραξικοπηματιών ή της προηγούμενης εκλεγμένης κυβέρνησης. Θα γνωρίζετε ότι κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει διάκριση μεταξύ μπανάνας ε, παραγωγής fair trade και μπανάνας παραγωγής ε, με φιλικές προς, τις, προς το περιβάλλον μεθόδους έναντι των μπανανών που παράγονται από πολυεθνικές. Και είπαμε να υπάρχει διαφοροποίηση του καθεστώτος ε, ως προς παραγωγούς μπανάνας ε, θεμητού και φιλικό προς το περιβάλλον εμπορίου. Ποια είναι η θέση σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι σημαντική αυτή η συμφωνία και ξεφύγαμε από τρεις ε, μεγάλες πολυεθνικές ε, και τις χώρες της Κεντρικής ε, Αμερικής και τα λοιπά. Ξεφύγαμε έτσι από μια διένεξη και θα ήθελα να ξέρω σύμφωνα με την Επιτροπή της Εκτιμήσεις της πώς έχει κατάσταση των μεριδίων αγόρας στην ευρωπαϊκή Πανταγορά για την μπανάνα από τις χώρες ΑΚΕ και σε διάφορες περιοχές ε, ε, Καναρία νησιά κλπ και που θα έχουν αυτό το νέο, τη νέα ποσόστοση γιατί κύριε Μπανάνα αυτή έχει την ε, το μεγαλύτερο μερίδιο. Τι θα γίνει, θα παραμείνουμε σε μια ενδιάμεση φάση για τους χώρους ΑΚΕ και για την μπανάνα των άλλων περιφέρων που είπαμε στην αρχή και τώρα ακόμα για τα 200 εκατομμύρια δεν θα επανέλθω αυτά που είπε ο Ζεντού και ο διπλανός μου συνάδελφος αλλά πώς ξέρουμε ότι είναι εντάξει το ποσό για αυτή τη μεταβατική περίοδο και αν κατανοράμε τελικά ότι δεν μας στάνει τι κάνουμε τότε, τι προτείνετε εσείς να γίνει και ακόμα σχετικά με τη διαδικασία που εσείς ο ίδιος δείξατε και ζητήσατε το Κοινοβούλιο του Ευρωπαϊκών να δώσει το πράσινο φως για την εφαρμογή την προσωρινή πριν τη σύμφωνη γνώμη ακριβώς σε τελική φάση, την τελική. Πεστε μας παρακαλούμε γιατί μας λέτε ότι εντάξει δεν θα είναι κάτι που δεν θα αλλάζει από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο δεν θα προσφέρει αυτή τη σύμφωνη γνώμη θα μπορέσει κανείς να επανέλθει να αλλάξει αυτή την προσωρινή εφαρμογή. Αλλά τι γίνεται όμως σε διεθνές επίπεδο. Ναι εντάξει υπάρχει μια διάθεση να έχουμε αυτό το καινούριο πράγμα στην αρχή να πούμε ναι και μετά να πούμε ότι α, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας. Θα πρέπει να δούμε ίσως είναι νωρίς για να έχουμε παρόμοιε δεσμευτικέ νομικά αποφάσει, αλλά είναι ένα θέμα που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Θα πρέπει να δούμε και έναν δρόμο εξόδου. Θα πρέπει να τον βρούμε από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο πει ότι υπάρχουν λόγοι να μην πει ναι, α πούμε, συμφωνή γνώμη. Τότε γιατί να πούμε εμεί ναι, πριν να πούμε το οριστικό του ναι. Και εδώ, χωρί να θυγούν και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και μετά και από αυτά που έχουμε βάσει το συνδίκη τη Αγώνα, να μην θίξουμε τα δικαιώματα τη αρμόδια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε την σύμφωνη γνώμη. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Μάτσο, αλλά από ό,τι ξέρω δεν είναι μέλος της Επιτροπής μας. Παρ' όλα αυτά μπορώ να του δώσω το λόγο αρκεί να είναι σύντομος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι φάνηκε καθαρά ότι προσφέρει ηρεμία και κυρίως στην Επιτροπή. Αλλά ο Πάλος Αλφα το είπε, δεν είναι όμως θετική συμφωνία. Για τους παραγωγούς δεν είναι θετική, τους κοινοτικούς. Ε, είναι εκείνοι που παράγουν εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα ήταν καλή συμφωνία αν δεν είχαμε αντισταθμιστικά μέτρα από πλευρά τη Επιτροπή και αυτό για του παραγωγού του κοινοτικού. Εντάξει, το να και, και οι Λετροαμερικάνοι είναι ικανοποιημένοι, αλλά οι κοινοτικοί παραγωγοί τι κάνουν, δεν είναι ικανοποιημένοι. Παραγωγοί που ζουν ακριβώ από αυτέ τι φοιτητικέ εκτολέψει του με το 76, με 176% και έχουν έχουν, 230 ε, ευρώ τον τόνο 176 ακριβώς είναι οι δασμοί. 148 εκεί παίρνουν ε, και ο ορίζοντα πάει προς τα 140. Αυτό επηρεάζει τα πράγματα εδώ το 2010 για τους κοινοτικού παραγωγούς ε, και τι γίνεται με τους μεγάλους διανομή που κάθε χρόνο εργάζονται ακριβώ και ήδη ζήτησαν ε, για το 2010 0,50 καταστά να μειωθεί η τιμή και για να πάμε από τα 186 στα 100 40 ευρώ, 180 ευρώ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, όλα αυτά η Επιτροπή υιοθέτησε μια συμφωνία για τα μέτρα βάσει σε ιστορικούς αριθμούς 2000-2005, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ακριβώς η Επιτροπή να βοηθάει έτσι, διακόπτει ο Πρόεδρος, κάτι που θα κοστίσει ακριβά στο μέλλον και εγώ είμαι καθαρά υπέρ αυτής της τεχνικής συνάντησης που προτείνει ο Πρόεδρος κ. Σόριβαν νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα. Θα ήθελα να στεριστώ και εγώ αυτές τις ερωτήσεις των Ισπανών ε, συναδέλφων για τις συνέπειες ε, που θα έχουν οι διατάξεις αυτές ε, στους κοινοτικούς παραγωγούς. μεταξύ άλλων στους παραγωγούς των Αζωρών, της Μαδέρας, των Καναρίων. υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις? Όχι, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σάλιβαν γιατί τέθηκε πληθώρα ερωτήσεων και έχουμε ελάχιστο χρόνο. Άντε, 7 λεπτά κύριε Σάλιβαν. Άντε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Καταρχήν, να απαντήσω στα ερωτήματα του κ. Ρίφ και Ντεζίρ ε, για αυτά τα σταθμιστικά μέτρα για τις χώρες ΑΚΕ. Εντάξει, λύθηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Κύριε Ρίφ, εσείς ρωτήσατε για την ε, εφαρμογή αυτού του, κανονισμού, αυτού του μέτρου του αντισταθμιστικού σε, στα θέματα της συναπόφασης σας δοθεί. Εδώ λοιπόν ε, ήδη ακούσαμε σήμερα πράγματα ανάμεσα στους συναδέλφους σας. Ναι, ναι, συγγνώμη, ήταν ε, του Προέδρου το μικρόφωνο ανοιχτό και όχι το δικό μου, γι' αυτό δεν ακουγόμουν. Καλά. Λοιπόν, ε, για το μηχανισμό προσαρμογής, ε, η απόφαση, ε, όλα αυτά θα γίνουν, θα δοθούν μέσω της συναπόφασης. Με, ζει με το Συμβούλιο θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο για τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος αυτού. Α το πω και μάλιστα ειλικρινά ότι δεν είμαι εμπειρογνώμων πάνω σε αυτές τις λεπτομέρειες που ιδιαίτερα συζητήθηκαν εδώ στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης με τους συναδέλφους ε, το χρόνο και αλλά κάτι ακόμα θα το ελέγξω συγχωρέστε με να δούμε αυτή τη βοήθεια που ενδεχόμενα θα είναι για όλες τις χώρες που παράγουν ε, μπανάνα αλλά σύμφωνα με κριτήρια που θα ζυγιστούν όλα αυτά θα ισχύσουν άλογα με το τι γίνεται στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας για τρία χρόνια ακόμα, κανονικά μέχρι το 2013, όχι πέρα από το 2013, είμαστε πέρα από τις δημοσιογραφικές προοπτικές και υπάρχει μια ρήτρα έτσι κάπως που λέει με το 2013 θα τα μελετήσουμε τα πράγματα ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα πετύχουμε μόνο για τους παραγούς, όχι ίσως και για την όλη δημιουργία υποδομή έχει να κάνει με τον ανταγωνιστικό τομέα λοιπόν και μια βελτίωση λιμένων πολλά και διάφορα, πολλά μέτρα μπορούν θεωρητικά να εφαρμοστούν ανάλογα με την μορφή δράσης. Εδώ στην τεχνική συνάντηση αυτή θα μπορούσε να παραστεί και από Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ένας συνάδελφος για να μας το αναλύσει λεπτομερέστερα. Αυτό που συζητήσαμε ήδη και με τις χώρες ΑΚΕ, αλλά παραλαμβάνω όλα αυτά θα σας δοθούν στα πλαίσια της υιοθέτησης των λεπτομεριών σε συναπόφαση από το Κοινοβούλιο λοιπόν. για τον κύριο Ζαντό, εντάξει, ναι, θετικό, θα σας δώσω τα στοιχεία αυτά, δεν τα θυμάμαι τώρα, από μνήμης ε, είναι κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, ε, θα σας τα πούμε όλα αυτά επισήμως ε, και με λεπτομερέστερα και μάλιστα γραπτός όπως το ζητήσατε. Για το θέμα της στάσης των χωρών και κύριε Χιγίνης. Το είπα και άλλοτε ότι το δέχτηκαν. Όχι με ενθουσιασμό, γιατί θα προτιμούσαν το στάτο κουβό φυσικά. Είναι σαφές. Αλλά αντιλήσαν πλήρως ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραμείνει το στάτο κουβό. Και για τους νομικούς λόγους των αποφάσεων του ΠΟΕ, αλλά και εξαιτία των διαπραγματευτικών δυσκολιών που είχαμε στα πλαίσια της DDA. Αντιλήφθησαν λοιπόν ότι αν επέμεναν η παραγωγή ΜΕΚ της Λατινικής Αμερικής κάτι που δεν είναι και παράλογο ότι οι μπανάνες θα είχαν ε, υποστεί περικοπή 80% ενώ τώρα μειώνονται κατά 30%. Οπότε δέχτηκαν ε, αυτή την λύση ως μη χείρον. Επίσης υπάρχει και μια διάβρωση των προτιμήσεων και έλαβαν και κάποια επιπλέον ε, οικονομική βοήθεια. Σίγουρα πολλοί πρόσωποι χωρονακέ θα ε, επικρίνουν αυτή την νέα ε, απόφαση, αλλά είχαν και εκείνοι συμφέρον να υλοποιηθεί συμφωνία γι' αυτό. Αλλιώ τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Για το θέμα της Ονδούρας, Η υπογραφή αφορούσε μια τεχνική προκαταρκτική συμφωνία και αυτό έγινε στη Γενέβη από τον πρέσβη ο πρέσβης ήταν ε, διορισμένος από την προηγούμενη κυβέρνηση και συνέχισε τη, την αποστολή του. Για το fair trade, το θεμητό εμπόριο, δεν θα ήταν εύκολο να βρούμε ε, τέτοια συμφωνία με τους παραγωγούς, γιατί θέλανε να καλυφθεί ολόκληρη η παραγωγή μπανάνας και δεν υπάρχει αποδεκτός ορισμός στο πω πώς θα γίνει η διάκριση μεταξύ των ε, δύο προϊόντων θεμητού εμπορίου και μαζικής παραγωγής. Εμείς προτιμούμε να ενημερώνουμε τον καταναλωτή ώστε να λάβει εμπεριστατωμένα μία απόφαση παρά να υποβάλουμε ε, άνοθεν και υποχρεωτικά μία διακριτική διαφοροποιημένη μεταχείριση. Επίσης ρωτήσατε για τα μερίδια αγοράς ε, ενώ θέλετε να σας δώσουμε αυτές τις στατιστικές. Διαθέτουμε ιδιαίτερα ακριβείς και παραδόξως μέχρι τώρα. Έστω και αν οι Ιταλογικοί δεσμοί μειώθηκαν υπέρ αυτών, τον ΜΕΚ ε, αυτά προκάλεσαν βέβαια και μια αντίδραση τότε των λατινοαμερικανικών χωρών ε, έστω και αν δεν, δεν αυτή η μείωση για τα προβλήματα στην αγορά. τέλο πάντων, τι να σα πω, είναι κάτι καστοριστικά ποσοστά, δεν είναι τεράστια και δεν θυμάμαι ακριβώ και τους αριθμού των γενετικών παραγωγών. Θα επανέλθω σε λίγο, αλλά σίγουρα θα σα δώσουμε τι σχετικέ στατιστικέ πάνω σε αυτό. Τώρα τι γίνεται, πώς επηρεάζει τα, μέρη αγορά, τα μέρη αγοράς ε, αυτή η συμφωνία. Να σας το πω και μας τα ειλικρινά, η αγορά μπανάνας ε, είναι από την παραγωγή μέχρι το να πάει στα μαγαζί είναι ε, παράξενη δομή. Τι να σας πω, τα μείωση των τελευταίων δασμών, πώς θα εκφραστούν όλα αυτά σε χαμηλότερες τιμές, σε μεγαλύτερα μέρη αγοράς. Τι να σας πω, είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Καμιά πολυοικονομική μέθοδος δεν υπάρχει να μας δείξει τι θα γίνει. Θα το δούμε αυτά σε καθημερινή πρακτική. Θα τα δούμε. Και τώρα για την προσωρινή συμφωνία. Νομίζω ότι αρκετά σαφής ήμουν ε, και είπα την επίσημη θέση ότι ε, υπογράψει το Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου μετά θα ακολουθήσει αυτή την πορεία και στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής υπάρχει και μια ρήτρα, ας το πούμε. Εντάξει, θα δούμε. Τι προβλέπετε αυτή τη συμφωνία με δύο στοιχεία τα οποία κανονικά θα ισχύσουν αμέσως. Παρά αυτά, μόλις έχουμε την υπογραφή Εντάξει, αυτό μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, θα το συζητήσουμε και να σας το πω ότι τα δύο αυτά στοιχεία επισήμως είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, εντάξει, γιατί κακό και άσχημο θα ήταν αν στην αρχή προχωρούσαμε και μετά πισαδρομούσαμε, προχωρούσαμε, Α, λοιπόν θα πρέπει να το δούμε, θα το εξετάσουμε αυτό για να δούμε πώς αυτά τα δύο στοιχεία θα μπορούσαν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Πάντως αυτό συνήθως χαρακτηρίζει ορισμένες συμφωνίες τεχνικού πολιτικού χαρακτήρα. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι και μεγάλε μεγάλες συμφωνίε τώρα έτσι ελευθέρων συναλλαγών, αλλά πάνω σε αυτά θα πείτε εσεί ε, ποια είναι η άποψή σα, θα δείτε ένα τρόπο ε, δουλειά ε, να κάνετε το χρέο σα και μπορεί να συνδυαστεί με τι όλε τι υποχρεώσει στα πλαίσια ε, διαπραγματεύσεων. Θα βρείτε μια λύση. Τέλος, για την κατάσταση των εγχώριων παραγωγών. Το μήνυμα ελήφθη. Δεν είναι βέβαια δική μου ευθύνη και αρμοδιότητα. Αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Πάντως παρατηρώ όμως ότι ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τους κοινοτικούς παραγωγούς είναι 279 εκατομμύρια το χρόνο. Κάτι που προστίθεται σε μια επιδότηση ανά επιφάνεια παραγωγής περίπου 10.000 ευρώ αναεκτάριο και αν κάνουμε σύγκριση με μια άλλη καλλιέργεια που είναι αδρά επιδοτούμενη, το βαμβάκι, που η βοήθεια είναι μεταξύ 252 με 271 ε, ευρώ το εκτάριο, διαπιστώνουμε ότι η επιδότηση για τις μπανάνες είναι σημαντική. Τώρα αν είναι αρκετή, δεν είναι δική μου ευθύνη να το κρίνω. Πάντως το θέμα της επιδότησης των εγχώριων παραγών μπανάνα σίγουρα θα συζητηθεί. Βέβαια, η θέση που λαμβάνει ο καθένα εξαρτάται από το κατά πόσο κατάγεται από χώρα που είναι παραγωγό μπανάνα ή όχι. Πάντω, εμεί ε, σε όλε τι φάσει ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ήδη δαψιλή υποστήριξη, ε, επιχορήγηση προ του χώρου παραγωγού. Άλλωστε η κατάσταση δεν αλλάζει αισθητά, είναι περισσότερο ε, διαμάχη μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και των χωρών που απολαμβάνουν καθεστώς μάλλον ευνομένο κράτους. Πάντως ε, και αυτό το θέμα της στήριξης των ε, τοπικών παραγωγών θα συζητηθεί. Πάντως εγώ είμαι στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και το ελέγχω αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμη συζήτηση, ήταν και προκαταρκτική συζήτηση, σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά θέματα. Η Επιτροπή μας θα εξετάσει αυτό το θέμα και θα σας ε, ξαναπροσκαλέσουμε εν καιρό για να εξετάσουμε τα διαδικαστικά ζητήματα που είναι επίσης σημαντικά. Αλλά ακόμη δεν το έχουμε συστήσει ούτε μεταξύ μας. Ωραία, η επόμενη μας συνεδρίαση προβλέπεται για τις 27 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ και καλό μεσημέρι.